Καλό απόγευμα σε όλους και όλες. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε λίγα άλλα εκλεκτά μέλη εδώ. Και έχουμε τη μεγάλη τιμή να έχουμε αυτή την τεράστια αίθουσα σήμερα. Ίσα ίσα σας βλέπω από αυτούς που είσαστε πίσω, στο πίσω μέρος αίθουσας. Ευχαριστώ για την έλευσή σας. Και πρωτού καλωσορίσω την Επίτροπο Ρέντινγκ, την Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, την κυρία Ρέντινγκ να σας ζητήσω να κρίνουμε την ημερησία διάταξη για την συνεδρίασή μας. Σας ευχαριστώ. Και απλώς <clears throat> να σας υπενθυμίσω ότι μεταδιδόμαστε στο διαδίκτυο. Χαιρετίζουμε αυτού που, αυτούς που μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο. Τα πρακτικά του Ιανουαρίου, 10 και 23-24 Ιανουαρίου είναι στο φάκελό σας και συνεχίζουμε την πατροπαράδοτη διαδικασία. Αν δεν υπάρξει αντίρρηση, η οποία θα διατυπωθεί μέχρι το τέλο τη συνεδρία, θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί. Περνάω λοιπόν στο κύριο θέμα τη σημερινή συνεδρίαση, που είναι η ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Ρέντινγκ, που είναι υπεύθυνη για θέματα δικαιοσύνη, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ηθαγένεια. Έχουμε συνεργαστεί πολύ στενά με την κυρία Ρέντινγκ στην Επιτροπή μας και στα πλαίσια της τρέχουσας θητείας και στο παρελθόν που ήταν αρμόδια για την κοινωνία της πληροφορίας και τα ΜΜΕ. Είναι ιδιαίτερα γνωστή λοιπόν σε όλους μας και είναι ένα άτομο το οποίο πάντα είναι πρόθυμο να έχει συζητήσεις με το Κοινοβούλιο. Κάναμε ένα γεύμα μαζί της την προηγούμενη εβδομάδα παρουσία των συντονιστών των πολιτικών ομάδων. Όλα αυτά ήταν πολύ χρήσιμα για να κατανοήσουμε τη μελλοντική στρατηγική της Κομισιόν και θα ακούσετε και περισσότερα σχετικά σήμερα. Θα προσκαλέσω λοιπόν την κυρία Ρέντινγκ να παρουσιάσει το μελλοντικό της πρόγραμμα εργασίας. Όλα αυτά εγγράφονται στο διαφθορμένο διάλογο που διενεργούμε μαζί με την Κομισιόν. Έχουμε πολλές ανεπίσημες επαφές μαζί σας και με την, τις υπηρεσίες σας. Τώρα όμως έχουμε αυτή την επίσημη ανταλλαγή απόψεων για να γνωρίσουμε ποια είναι τα σχέδιά σας, ιδίως ό,τι αφορά το κεκτημένο στα θέματα καταναλωτών που αντιμετωπίζει η κυρία Ρέντινγκ γιατί ως Επιτροπή θέλουμε και εμείς Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς θέλουμε να δώσουμε και εμείς συνέχεια μαζί με την Κομισιόν στα θέματα αυτά στο υπόλοιπο τμήμα της θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι απεριόριστος ο χρόνος αυτός βέβαια και γι' αυτό θέλουμε να εστιάσουμε ώστε να τον καλύτερα την προσοχή μας στα πιο σημαντικά θέματα Μπορώ λοιπόν τώρα μετά από όλα αυτά να ζητήσω από την κυρία Ρέντινγκ να λάβει το λόγο ενώπιον της Επιτροπής μας και ελπίζω ότι θα έχετε και κάποια σχόλια και ερωτήματα. Η κυρία Γάδοβης έχει ήδη ζητήσει το λόγο και όποιος άλλος θέλει να λάβει το λόγο το καταγράφω. Έχετε το λόγο λοιπόν κυρία Ρέντινγκ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, έντιμα μέλη της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που απευθύνατε να λάβω το λόγο ενώπιόν σας να στραφώ κατευθείαν στα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν την Επιτροπή σας και σας είναι προσφυλή τα ζητήματα προστασίας των καταναλωτών και η νομοθεσία για τους καταναλωτές. Το Μάιο του 2012, όπως ξέρετε, η Κομισιόν έχει εγκρίνει, ενέκρινε μάλλον ένα φιλόδοξο σχέδιο για την πολιτική καταναλωτών από τώρα έως το 2020. Είναι η ατζέντα των καταναλωτών και αυτό όχι μονάχα μετά από τις εκκλήσεις της δικής σας Επιτροπής και της έκθεσης του 2011 που ήταν μια σημαντική ε, έκθεση που απετέλεσε και έναυσμα για την εργασία μας. Το ερώτημα που μας ενδιαφέρει είναι το πώς θα προχωρήσουμε για τα θέματα των καταναλωτών, πώς θα εξασφαλίσουμε ότι οι καταναλωτές μπορούν να επιλέγουν εν γνώση των πραγμάτων και υποστηρίζοντας τον ανταγωνισμό ο οποίος οδηγεί σε μια ανάπτυξη η οποία είναι πιο αποδοτική σε σχέση με την χρήση των πόρων. Ο στόχος μας στην πολιτική καταναλωτών επομένως είναι να εξασφαλίσουμε την καλύτερη εφαρμογή των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Μόνο στην περίπτωση που είναι <clears throat> δυνατόν να ισχύουν και να εξασφαλίζονται τα δικαιώματα των καταναλωτών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν γίνει σαφές ότι οι ασυνείδητοι έμποροι και αυτοί οι οποίοι προβαίνουν σε αθέμητο ανταγωνισμό θα υφίστανται κυρώσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο έτσι μπορούμε να προωθήσουμε την εμπιστοσύνη σε θέματα όπως η ψηφιακή επανάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δίνει περισσότερες δυνατότητες για αγοραπολισία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δυστυχώς δίνει και λαδί σε περισσότερες αθέμητες ε, συναλλαγές από εμπόρους χωρίς πραγματική επαγγελματική συνείδηση. Στις επερχόμενες συζητήσεις μας θα δούμε περισσότερο και πώς θα μπορέσει να γίνει αυτή η καλύτερη εφαρμογή του καταναλωτικού δικαίου. Η οδηγία λοιπόν για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Βρισκόμαστε στη φάση υλοποίησης και η οδηγία αυτή είναι σημαντική γιατί θα αποδώσει περισσότερα δικαιώματα στους καταναλωτές η περίοδος απόσυρσης των 14 ημερών, η κατάργηση των υπερβολικών επιβολών τελών μέσω πιστοτικών καρτών, όλα αυτά είναι σημαντικά στοιχεία για τους καταναλωτές και γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η εφαρμογή αυτών των κανόνων στην πράξη θα μπορέσει να γίνει με τον πρέποντα τρόπο και θέλουμε να δώσουμε και την απαραίτητη κατεύθυνση όταν αυτό είναι απαραίτητο προς τα κράτη-μέλη, κυρίως με εργαστήρια και ατελιέ όπου συζητείται η συγκεκριμένη υλοποίηση στο εθνικό δίκαιο των θεμάτων αυτών. Βέβαια, ένα βασικό πρόβλημα είναι η γνώση των δικαιωμάτων τους από την πλευρά των καταναλωτών. Αν δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, αυτά τα δικαιώματα είναι ατελέσφορα. για αυτό τον λόγο. Στο πέρας του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών, Εγώ εντυπωσιάστηκα που δεν υπήρξαν πολλά ερωτήματα για τα δικαιώματα των καταναλωτών τα οποία να γερθούν μέσα σε αυτό το έτος. Γι' αυτό είναι απαραίτητο κατά την άποψή μας να έχουμε μια εκσταθία συνειδητοποίηση των καταναλωτών ώστε να διευρυνθεί η γνώση των καταναλωτών σε σχέση με τα δικαιώματά τους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις και οι οργανώσεις των καταναλωτών θα εμπλέκονται πλήρως σε αυτή την εκσταθία και με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και τη μεγαλύτερη διάδοση αυτών των γνώσεων. Για τα θέματα της ψηφιακής ατζέντα. Ξέρετε ότι η ατζέντα για τους καταναλωτές περιλαμβάνει και δράσεις για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε ψηφιακά προϊόντα, αυτά τα οποία πουλούνται επιγραμμικά ή μέσω κινητών τερματικών συσκευών. Η νομοθεσία <clears throat> της, για τους καταναλωτές και οι αντίστοιχες πρόνοιες προβλέπουν διασφαλιστικές ρήτρες για τα προϊόντα τα οποία αγοράζονται με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή από το διαδίκτυο ή με κινητές συσκευές. Το θέμα είναι πόσο αποτελεσματική είναι η εφαρμογή αυτών των δικαιωμάτων. Επομένως, ο στόχος μας είναι να δημοσιεύσουμε κατευθυντήριες γραμμές για τις πληροφορίες οι οποίες πρέπει να δίνονται, να έχουμε ένα υπόδειγμα επιχειρηματικής συναλλαγής που να αναφέρει τις κύριες πληροφορίες οι οποίες πρέπει να υπάρχουν και επίσης να χρησιμοποιήσουμε δίκτυα όπως το CPC για να εξασφαλίσουμε την καλύτερη υλοποίηση και αστυνόμευση της εφαρμογής αυτών των δικαιωμάτων. Όλα αυτά με φέρνουν σε ένα σημείο της ημερήσιας διάταξης που σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, η ψηφιακή ενιαία αγορά και εδώ υπάρχουν δύο κέρυε προτάσεις. Καταρχήν το, ευρωπαϊκό, το κοινό ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο ή καλύτερα δίκαιο για τις πωλήσει. Εγώ αποδίδω μεγάλη σημασία στα θέματα αυτά γιατί είναι σημαντικό σε μια περίοδο ισχνών αγελάδων να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα κερδοφορίας για τους εμπόρους αλλά και εξοικονόμησης για τους καταναλωτές. Επομένως, η κοινή νομοθεσία για τις πωλήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ισχυροποιήσει και την προστασία των καταναλωτών σε σχέση με τον προηγούμενο κεκτημένο <clears throat> της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα προχωρήσει ακόμα πέραν των περισσότερων εθνικών νομοθεσιών για τα θέματα αυτά. Το ελάχιστο όμως το οποίο πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι το σημερινό και εκτιμένο. Είναι το ελάχιστο κατόφλιο στο οποίο πρέπει να βρεθούμε όλοι. Θέλουμε να προχωρήσουμε όμως ακόμα περισσότερο και θέλουμε να δημιουργήσουμε και περισσότερες δυνατότητες στην ψηφιακή ενιαία αγορά που θα είναι ένας από τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης, θα αυξήσει την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή αγορά, ώστε οι καταναλωτές και οι έμποροι να μπορούν να έχουν μεγαλύτερη αμοιβαία εμπιστοσύνη όταν γίνονται αγοραπολισίες ψηφιακών προϊόντων, ακόμα και αυτών που θα βρίσκονται αύριο στο υπολογιστικό νέφος. Και εμείς ε, περιμένουμε και από εσά να ελέγξετε και να αξιολογήσετε αυτές τις προτάσεις και περιμένουμε τις προτάσεις των συνεισηγητών σας για τα θέματα αυτά, ώστε να μπορέσει η νομοθεσία αυτή να καρποφορήσει ήδη μέσα στο τρέχον έτος και η Κομισιόν φυσικά οικοθενοείται ότι είναι έτοιμη να παίξει ένα διαμεσολαβητικό και διευκολυντικό ρόλο εναντί του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να ευοδοθούν οι προσπάθειες αυτές. Γνωρίζω επίσης ότι η Επιτροπή σας ενδιαφέρεται ιδιαίτερα στο να εξασφαλιστεί η καλύτερη ισορροπία μεταξύ των επιχειρηματικών ευκαιριών από τη μία πλευρά και της προστασίας των καταναλωτών από την άλλη πλευρά. Είμαι δεσμευμένη να εξασφαλίσω και να διατηρήσω αυτό το υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ώστε η νέα αυτή νομοθεσία να αποτελέσει μια ελκυστική λύση για τις επιχειρήσεις. Να κατανοήσουν λοιπόν και αυτοί ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και τους καταναλωτές. Και όσο μιλάμε για τον ψηφιακό χώρο, την ενιαία ψηφιακή αγορά, φυσικά θα εφαρμόζονται και οι νέοι κανόνες για την προστασία δεδομένων και θα έχουν ζωτική σημασία γιατί εξασφαλίζουν αυτό το οποίο και εσείς θέλετε να επιτύχετε στην Επιτροπή σας, την διεύρυνση της ενιαίας αγοράς και τη δημιουργία μιας πραγματικής ψηφιακής αγοράς και την εξασφάλιση παράλληλα της προστασίας των πολιτών και των καταναλωτών. Έχουμε επιτύχει θετική πρόοδο στα θέματα αυτά. Παρακολουθούμε τη συζήτηση μεταξύ των συνομοθετών, τις συζητήσεις και στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στην Ιρλανδική Προεδρία η οποία θέλει να προωθήσει αυτές τις διαπραγματεύσεις ώστε να υπάρξει συμφωνία τουλάχιστον σε μια γενική προσέγγιση μέχρι το τέλος της Ιρλανδικής Προεδρίας στο Συμβούλιο Εσωτερικών και Δικαστικών του Ιουνίου. Και είναι μεγάλη ικανοποίηση για μας το να γνωρίσουμε ότι υπάρχει μια σειρά από θέματα τα οποία την χάνουν γενική ομοφωνία σε σχέση πραγματικά χάρη για το αδρό περίγραμμα για την αρχιτεκτονική της μεταρρύθμισης. Αυτό γίνεται γενικά αποδεκτό ως συνενετικό στοιχείο. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η μεταρρύθμιση είναι πολύ σημαντική διότι μπορεί καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων να μείνει σαν μια διαπραγμάτευση που οδηγεί σε θετικό άθεσμα, σε μια κατάσταση που κερδίζουν όλοι. Αντί να υπάρχει κατακαιρματισμός σε 27 ή 28 χώρους κανόνων και έγκριση το να υπάρχει μονάχα μια διαδικασία έγκρισης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγχρόνως όταν υπάρχει ενίσχυση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις συνθήκες και από τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για όλους τους πολίτες μας σε ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο προχωράει θετικά και γι' αυτό θα είμαι ευγνώμων σε όλους αυτούς οι οποίοι θα μπορέσουν να βοηθήσουν να εξευρεθεί μια θετική για όλους λύση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να βρει τρόπους ανταπόκρισης στις αλλαγές οι οποίες έχουν υπάρξει στην κοινωνία μας τα τελευταία χρόνια. Ξέρετε ότι οι ομαδικές μετακινήσεις από τότε που δημιουργήθηκαν και τα οργανωμένα ταξίδια πάρα πολλοί Ευρωπαίοι ε, αγόραζαν στα πρακτορία ε, τα ταξίδια τους, ενώ τώρα το κάνουν αυτό στο ε, διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός πελατών δεν ε, περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις της προηγούμενης οδηγίας. Εγώ άκουσα τις απόψεις της βιομηχανίας του τουρισμού σχετικά με τις προτάσεις για την αλλαγή των ρυθμίσεων σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια. Άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά τις ανησυχίες των καταναλωτών και έχουμε τρεις επιλογές. Η πρώτη είναι να εξυγχρονίσουμε την ισχύουσα νομοθεσία. Η δεύτερη είναι να την αφήσουμε ως έχει. Και η τρίτη επιλογή είναι να την διαγράψουμε πλήρως. Εγώ παρακολούθησα και την τελευταία διαβούλευση ανάμεσα στους εμπλεκομένους και στο τέλος της Άνοιξης εμείς θα πάρουμε μία απόφαση σχετικά με τις ρυθμίσεις αυτές. και θα σας ενημερώσουμε έτσι ώστε και εσείς να μπορέσετε να συμμετέχετε στο τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ δεν έχω αποφασίσει ακόμα τι θα κάνω, λέει η Επίτροπος. Προς το παρόν ακούω, αλλά ε, θα ήθελα και από πλευρά σας προτάσεις πριν από την άνοιξη του 2014, Επίτροπος. Τώρα για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές και την οδηγία που τις αφορά. Αυτά εντάσσονται στην ημερήσια διάταξη που ασχολείται με τους καταναλωτές. Τον Μάρτιο φέτος θα ξεκινήσουμε με μια ανακοίνωση και μια έκθεση σχετικά με την πρώτη αξιολόγηση της εφαρμογής συγκεκριμένη οδηγίας. Η επόμενη φάση είναι μια θα έλεγα επισκόπηση της εφαρμογής της οδηγίας αυτής και η έκθεση θα αφορά κάποια πολύ συγκεκριμένα θέματα όπως η εφαρμογή της συγκεκριμένη οδηγίας στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, σε ακίνητα και στην προώθηση πωλήσεων. Τα πρώτα χρόνια εμπειρίας της εφαρμογής της οδηγίας αυτές για τις αθέματες εμπορικές πρακτικές μας έδειξε ότι μπορεί να ωφελήσει και τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Και ως προς αυτό λοιπόν έχει συνεισφέρει στη βελτίωση της προστασίας του καταναλωτή στα κράτη-μέλη, προωθώντας και τα συμφέροντα των επιχειρήσεων και προστατεύοντας τις επιχειρήσεις από ανταγωνιστές που δεν σέβονται τον κανονισμό. Πάντως θα θέλαμε εμείς η οδηγία να αποδώσει ακόμα περισσότερο στον τομέα της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς και το θέμα το οποίο τίθεται ο συνήθως είναι η σωστή εφαρμογή. Συγκριτικές διαφημίσεις, παραπλανητικές διαφημίσεις. Τι γίνεται με την οδηγία αυτή. Αυτό δεν αφορά μόνο τους καταναλωτές αλλά και τις επιχειρήσεις. Και οι επιχειρήσεις χρήζουν προστασίας από τέτοιου είδους πρακτικές. Και αναφέρομαι εγώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες πέφτουν θύματα τέτοιων διαφημίσεων ιδιαίτερα σε διασύνοριακές συναλλαγές. Η οδηγία που ισχύει παρέχει ένα πλαίσιο προστασίας. Υπάρχουν όμως ενδείξεις ότι χρήζει εξυγχρονισμού. Θα πρέπει να γίνει πιο αυστηρή. Εμείς ήδη δημοσιεύσαμε μία ανακοίνωση και εγώ θα καταθέσω μία νομοθετική πρόταση κατά τη διάρκεια του 2013. Δύο θα είναι οι βασικές μας προτεραιότητες. Πρώτον, οι κανόνες που απαγορεύουν ορισμένες τέτοιες εμπορικές πρακτικές να είναι πιο σωστά προσαρμοσμένοι στη σημερινή πραγματικότητα και δεύτερον να ενισχύσουμε την ενίσχυση της προσπάθειας καταπολέμησης αθέμητων πρακτικών. Νομίζω ότι εδώ μπορούμε να συνεισφέρουμε και να βοηθήσουμε μέσω της μεταρρύθμισης, της ρύθμισης. Ένα άλλο στοιχείο, το οποίο σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, κύριος Μάγερ ασχολείται με θέματα νομικής συνδρομής σε διασυνοριακές συναλλαγές και διαφορές. Δεν έχει ρυθμιστεί το θέμα πλήρως, δεν έχει υπάρξει απόφαση ακόμα ενώ. Βασίζεται η προσπάθεια αυτή στην οδηγία του 2003 έτσι ώστε να μπορέσουν ε, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσουν τα μέτρα που τους παρέχει η δικαιοσύνη και σε άλλες χώρες μέλη. Έχουμε εντοπίσει ε, κάποια εμπόδια και κάποιες αδυναμίες στην εφαρμογή της οδηγίας επί τη βάση της έρευνας την οποία είχε υπογραμμίσει η έκθεσή μας. Εδώ έχουν γίνει προτάσεις και από σας σας ευχαριστώ για τις προτάσεις σας, τις οποίες αποστήλατε και στα κράτη-μέλη. Το θέμα είναι ε, ότι οι πολίτες δεν συνειδητοποιούν ότι έχουν δικαιώματα, δυστυχώς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επανέρχομαι σε αυτά τα οποία είπα. Απαιτείται να υπάρξει μια εκστρατεία πληροφόρησης. Ένα θέμα σημαντικό είναι η σωστή κατάρτιση των δικηγόρων, των νομικών. γιατί το θέμα εδώ δεν εμπλέκεται μόνο, δεν εμπλέκει μόνο τα δικαιώματα των καταναλωτών, αλλά και θέματα δικαιοσύνης γενικότερα. Οπότε προσπαθούμε και μέσα από τα προγράμματα που αφορούν τη δικαιοσύνη να βοηθήσουμε. Επίσης και με την προσπάθεια επίλυσης διαφορών με ένα λακτικό τρόπο. Είναι κάτι το οποίο και αυτό ενδιαφέρει τις σχέσεις καταναλωτών και επιχειρήσεων. Πολλές φορές για ρυθμίσεις τέτοιων διαφορών δεν απαιτείται η προσφυγή στα δικαστήρια. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ότι αυτές οι εναλλακτικέ ε, προσπάθειες λύσης των διαφορών είναι αξιόπιστες, η ενημέρωσή τους είναι σωστή, ε, εξετάζουμε σε αυτή τη φάση την ομοθεσία η οποία τώρα έχει αρχίσει να εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη και γι' αυτό στα πλαίσια μιας εκστρατείας πληροφόρησης θα πρέπει να ενημερώσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Να ξεπεράσουμε λίγο αν θέλετε ακόμα και αυτά τα οποία εσείς κάνετε και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα των πολιτών οι οποίοι πολλές φορές δεν γνωρίζουν ποια είναι η αρμόδια επιτροπή και ε, ζητούν από εμά το τι θα πρέπει να κάνουν. Well, thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω μία ολόκληρη σελίδα με τις σημειώσεις σχετικά με τα θέματα που θα ήθελα να αναφέρω. Πριν αρχίσουμε τη συζήτηση, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερος που θέσατε το θέμα για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του καταναλωτή και γενικά του πολίτη. Γιατί νομίζω ότι, όπως είπατε, σωστά είπατε μάλλον, οι μικρές επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται και τι ακριβώς προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και αυτό το έχουμε σημειώσει ιδιαίτερω στο πλαίσιο κάποιων συγκεκριμένων ε, project. Έχουμε πλέον ε, στην Γενική Διεύθυνση Αγοράς ε, ένα φυλάδιο για τα δικαιώματα του πολίτη στην εσωτερική αγορά. Θεωρώ ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα προωθήσουμε περαιτέρω και να εξετάσουμε και άλλα ζητήματα για ενδεχόμενες εκστρατείε. κάποια έκθεση πρωτοβουλίας ίσως για την πολιτική αυτή. Γιατί νομίζω ότι αυτό μας αφορά όλους μας. Τώρα, να ακούσουμε τι έχουν να πούν τα μέλη της Επιτροπής. Μέχρι τις 4 νομίζω έχετε ώρα. Σε ομάδες των τριών, λοιπόν, αν θα θέλετε να κάνετε συνοπτικές ερωτήσεις για να ξεκινήσει ο διάλογος. Γκάλο, Σενέλοβα και κυρία Ράπτη. Ο πρώτος γύρος. Uh, uh, Στο δεύτερο γύρο, κανείς άλλος. θέλει να πάρει το λόγο ο κύριος Ρόσφο, ο κύριος Σβάμπ. ως εισηγητής για την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών, ξέρω ότι σίγουρα θα θέλετε το λόγο. Μάλιστα, λοιπόν, τρεις γύρους ερωτήσεων ως τώρα. Merci, le Président. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για τις εξηγήσεις που μας δώσατε και σας ευχαριστώ για το γεγονός ότι μας υπενθυμίσατε ότι για την ανάπτυξη της ε, ψηφιακής ενιαίας αγοράς είναι απαραίτητο οι συμπολίτες μας, που τους αναφέρουμε βέβαια ως καταναλωτές σήμερα, θα πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στις συναλλαγές και εμπιστοσύνη στους φορείς με τους οποίους συναλλάσσονται. Εγώ ως εισηγήτρια στην νομική επιτροπή για τον κανονισμό που αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων παρακολουθώ αυτό το θέμα αλλά επίσης και ως Γαλλής και θα καταλάβετε γιατί με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα αυτό. Στην ε, περιοχή του Παρισιού στις 28 Φεβρουαρίου έλαβε χώρα ένα σεμινάριο διοργανωμένο από τη Γαλλική Σοσιαλιστική Κυβέρνηση σε σχέση με την ψηφιακή ατζέντα. Ο οδικός χάρτης ο οποίος δημοσιεύτηκε μετά από αυτό το σεμινάριο προέβλεπε ότι θα πρέπει να αναθεωρηθούν όλες αυτές οι ρήτρε προστασίες των πολιτών ώστε να απο... αποκομίσουν μεγαλύτερο επίπεδο προστασίας ιδίως για τα πιο ευάλωτα άτομα, για τους νέους κτλ. Αστυνομικές ε, δράσεις επίσης προβλεπόταν για να εξασφαλίσουν όλα αυτά τα στοιχεία. Όλα αυτά βέβαια ήταν ήδη στην οδηγία και τελικά εκφράστηκαν και συγκεκριμένα ορισμένες αμφιβολίες και ανησυχίες και αναφέρθηκε και το δικό σας όνομα κύριε Επίτροπε. Είπαν ορισμένοι ότι φοβούνται πάρα πολύ ότι από αυτό το νέο ευρωπαϊκό κανονισμό θα προκύψει μια ισοπαίδωση προς τα κάτω και ιδίως σε ό,τι αφορά την εναρμόνιση των κυρώσεων και αυτό θα μείωνε και την δύναμη των εθνικών αρχών στην επιβολή κυρώσεων. Όλα αυτά λοιπόν ήταν οι ανησυχίες και οι φόβοι που εκφράστηκαν από τη, από τη γαλλική κυβέρνηση πρόσφατα και εγώ έχω αυτή την ανησυχία που θέλω να σας μεταφέρω. Θα ήθελα να έχω τη δική σας άποψη σχετικά γιατί πιστεύω ότι κάθε κράτος ε, μέλος θα πρέπει να εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία και να κινητοποιηθεί για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτός ο κανονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ενδιαφέρουσες αυτές παρατηρήσεις που γίνονται σε σχετικά με τις συζητήσεις που γίνονται σε άλλες χώρες και νομίζω ότι δεν είναι η μοναδική η γαλλική κυβέρνηση που ασχολείται με τέτοια θέματα. Η κυρία Σενέλεβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κυρία Επίτροπε για την εισαγωγή. Θα μιλήσω αγγλικά αυτή τη φορά γιατί παίρνω το λόγο εξ ονόματος της κυρίας Γκέπχαρτ, ε, της συντονιστριάς μας που δεν μπορεί να είναι παρούσα σήμερα και είναι και συνηθιγήτρια σε ό,τι αφορά την έκθεση για το κοινό εμπορικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ξέρετε, εδώ και χρόνια θέλουμε να συμβάλλουμε στην καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και προσπαθούμε να βάζουμε τον, Ευρωπαϊκό, τον Ευρωπαίο πολίτη στο κέντρο της πολιτικής μας εργασίας. Η προτάση όμως για το Common European Sales Law δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων και η κριτική που ασκείται κατά της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ καλά, είναι πολύ καλά τεκμηριωμένη. Βασίζεται και μάλιστα στο health check, στο μελέτη αντικτύπου που έγινε από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τονίζουμε τα εξή στοιχεία. Καταρχά, τον υπολογισμό τον, του κόστου των σε σελίδε 13 και 14. Ο υπολογισμό αυτό ε, βασίζεται σε δύο μη αντιπροσωπευτικέ μελέτε και άνω του ίμιση των εμπορευομένων δεν έδωσαν τέτοιες αξιόπιστες ε, πληροφορίες σε σχέση με το κόστος συναλλαγής. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να βασιστούμε στις, στους υπολογισμούς αυτούς που έγιναν από τους εμπορευόμενους ουσιαστικά. Σε ό,τι αφορά τώρα τα εμπόδια για το διασυνοριακό εμπόριο μεταξύ των επιχειρήσεων. Αυτό είναι πολύ υπερτιμημένο μετά την εφαρμογή του κοινού ε, εμπορικού δικαίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει να μειωθούν οι τιμές σε επίπεδο 0,04 έως 0,07%. Κατά δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίστηκε σε κάποιες αδικαιολόγητες ε, εικασίες για την αύξηση, για παράδειγμα, της βάσης των πελατών, μόνο επειδή θεωρείτε ότι θα υπάρχει μια ε, ετικέτα ποιότητας. Είναι πραγματικά πολύ ενοχλητικό πόσο αναξιόπιστα είναι τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η μελέτη αντικτύπου. Δύο ερωτήσει τώρα. Πώς αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή αυτά τα πορίσματα του Health Check του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα υπάρξει αντίκτυπος σημαντικός στη μετέπειτα δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ό,τι αφορά αυτό το κοινό ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο. Ευχαριστώ πολύ. Σημειώνουμε λοιπόν τα σημεία αυτά που δείξατε και στο γύρο αυτό σίγουρα θα συζητηθούν και τα θέματα αυτά πιο πολύ. Η κυρία Ράπτη όμως τώρα έχει το λόγο τελευταία σε αυτό το γύρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κυρία Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Ρέντινγκ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Ρέντινγκ, το ξαναλέω για τη μετάφραση. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ σήμερα. Άκουσα με πολύ προσοχή την ομιλία σας και ομολογώ ότι ε, με έκανε να ελπίζω ότι θα ανταποκριθείτε στις προκλήσεις που υπάρχουν μπροστά σας για να γίνει καλύτερη η ζωή των καταναλωτών. Συνήθως κάθε φορά που έρχεστε στην Επιτροπή έρχονται στο μυαλό μου δύο πράγματα. Το ένα είναι η οδηγία για το roaming και το άλλο είναι οι αγώνες που έχετε κάνει και συνεχίζετε πάντα να κάνετε για το ζήτημα της ισότητας των φύλων Έχουμε και την ημέρα της γυναίκας σε μερικές μέρες. Αυτό λοιπόν με κάνει να ελπίζω ότι θα ανταποκριθείτε και στις πολύ ισχυρές προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας τώρα. Στην, επόμενη, στην ερχόμενη ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ψηφιστεί ε, το Alternative Dispute Resolution Mechanism που όπως είπατε και στην εισήγησή σας είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, αυτό μας κάνει να ελπίζουμε ότι θα βελτιωθεί η ζωή των καταναλωτών. Ωστόσο υπάρχουν πάντα οι περιπτώσεις σύμφωνα με τις οποίες δεν μπορεί να βρεθεί λύση για τα προβλήματα των καταναλωτών μέσω του ADR. Και εκεί ακριβώς έρχονται να τοποθετηθούν οι collective redress θυμίζω ότι είχε γίνει εδώ και δύο χρόνια είχε ξεκινήσει μια διαβούλευση με πρωτοβουλία της Κομισιόν στην οποία δόθηκαν 18.000 απαντήσεις. Σύμφωνα με τις απαντήσεις αυτές και έτσι όπως αναφέρεται σε μια έκθεση της Κομισιόν υπάρχει η προτροπή από την πλευρά των καταναλωτών η προτροπή από την πλευρά αυτών που απάντησαν να πάρει η κομισιόν νομοθετικά μέτρα. το ίδιο ακριβώς ζητάει και το κοινοβούλιο με ένα συγκεκριμένο ψήφισμα που είχε στις 2 φεβρουαρίου του 2012. Ε, περιμέναμε ότι μέσα στο 2012 θα βλέπαμε αυτά τα νομικά μέτρα για το collective redress. Ε, δεν το είδαμε. Ε, θέλω να ξέρω πραγματικά τι θα περιμένουν για αυτό το θέμα οι καταναλωτές και το λέω ε, γιατί έτσι όπως τοποθετηθήκατε για διάφορα ζητήματα όπως τα ταξίδια όπως οι διασυνοριακές συναλλαγές όπως η ε, τεχνολογία που αρχίζει ε, κάθε καταναλωτής μόνος του να συναλλάσσεται στο διαδίκτυο το είπατε κι εσείς δημιουργεί ένα άλλο περιβάλλον και εκεί νομίζω ότι το collective redress είναι αυτό που θα δώσει ασφάλεια στον καταναλωτή σε σχέση ιδιαίτερα με το διασυνοριακό εμπόριο. Θα περιμένω έτσι με ανυπομονησία την απάντησή σας. Ευχαριστώ πολύ. Επίτροπε, θα θέλετε να απαντήσετε στα τρία αυτά ερωτήματα και μετά θα ακούσουμε άλλες τρεις ερωτήσεις. Uh, uh, Η πρώτη ερώτηση για την προστασία των δεδομένων και τη μεταρρύθμιση των μέτρων προστασίας. Όπως ήδη είπα, εδώ έχουμε δύο σοβαρές επιπτώσεις. Η πρώτη είναι εμπορικού τύπου. γιατί από τη μία δεν θα υπάρχουν 27 νομοθετικές ρυθμίσεις αντιτιθέμενες, αλλά μία ενιαία για το σύνολο της Υπήρου. Αυτό σημαίνει ότι θα εξοικονομήσουμε 2,3 δις ε, για τις επιχειρήσεις σε αιτήσια βάση. Πρόκειται λοιπόν για ένα μέτρο που ανοίγει αγορές. Θα μπορούσε βέβαια να πει κανείς στα πλαίσια αυτής της λογικής ότι αν υπάρχει ένας κανόνας για μία ήπειρο, τότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει και ένα συνολικός ε, εποπτικός οργανισμός. Εγώ είπα ότι δεν χρειάζεται αυτό. Και το είπα γιατί οι εθνικές εποπτικές αρχές γνωρίζουν τις αγορές τους, γνωρίζουν τους παίκτες τους, γνωρίζουν τους πολίτες τους. Και γι' αυτό ακριβώς εγώ αποφάσισα να έχω μια θηρίδα ενιαία one stop η οποία να δίδει περισσότερες δυνατότητες στις, εθνικές, στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές στο έδαφος τους. Αλλά θα πρέπει οι αρχές αυτές να εφαρμόζουν τους ιδίους κανόνες και ταυτόχρονα οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες και από τις επιχειρήσεις και από τις κυβερνήσεις και θα πρέπει επίσης να είναι επαρκώς εξοπλισμένες οι εποπτικές υπηρεσίες για να ασκούν τα καθήκοντά τους. Μιλάμε λοιπόν για την ενίσχυση των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και ως προς αυτό έχουμε εμπνευστεί από τα σωστά παραδείγματα και η ΚΝΙΛ η υπηρεσία αυτή είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Δεν είναι τυχαίο γιατί το άρθρο 29 της ομάδας εργασίας που περιλαμβάνει <clears throat> όλες τις ρυθμιστικές αρχές ζήτησε από την ΚΝΙΛ να προχωρήσει στην ανάλυση των τελευταίων προβλημάτων που έχουν σημειωθεί από πλευρά των επιχειρήσεων. Συνεπώς λοιπόν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ακόμα και σήμερα θα έλεγα ασκούν τις αρμοδιότητές τους όπως προβλέπονται από τον κανονισμό. Ήδη πριν δηλαδή τεθεί σε λειτουργία ο κανονισμός εφαρμόζουν τη διαδικασία του One Stop Shop. Αυτό είναι κάτι το οποίο εξυπηρετεί και τα συμφέροντα των εργαζομένων αλλά εξυπηρετεί και τις επιχειρήσεις και τον τρόπο που τις αντιμετωπίζουμε. Κάθε ρυθμιστική αρχή ασχολείται και ελέγχει τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν σεβαστεί τις εθνικές νομοθεσίες, τις εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις και επιβάλλουν κυρώσεις. Κάποιες εποπτικές αρχές δεν έχουν το δικαίωμα αυτό και η μέγιστη ποινή η οποία μπορεί να επιβληθεί είναι γύρω στις 600.000 ευρώ. Υπάρχουν όμως τρεις ρυθμιστικές αρχές που μπορούν να επιβάλλουν τέτοια πρόστιμα. Για κάποιες από τις επιχειρήσεις μας αυτές το ποσό αυτό είναι χαρτζηλίκι βέβαια. Και γι' αυτό προτείνω όλες οι ρυθμιστικές αρχές να μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμα που να φτάνει το 2% του συνολικού παγκόσμιου τζίρου κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων. Και η πρόσοδος αυτή θα βελτιώσει ε, και τις δυνατότητες που έχουν οι ρυθμιστικές αρχές, θα έχουν όλα τα μέσα τα οποία έχουν ανάγκη και έτσι θα αναλάβουν δράση αν χρειαστεί, ενώ πραγματικά δεν θα χρειάζεται και οι επιχειρήσεις θα γνωρίζουν ποιο θα είναι το τίμημα του μη σεβασμού του νόμου. Λοιπόν, ο κανονισμός αυτός με ισχυρό τρόπο ενισχύει τις δυνατότητες των ρυθμιστικών αρχών να εφαρμόσουν τις κοινέ νομοθετικές ευρωπαϊκές ρυθμίσεις και δεν είναι μια εξίσωση προς τα κάτω αλλά προς τα άνω. Γιατί ακριβώς έχουμε χρησιμοποιήσει τις καλύτερες των αρχών αυτών και τα επίπεδα τα οποία εφαρμόζουν και τα έχουμε καταστήσει ακόμα πιο αυστηρά και υψηλά. Είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει όλες τις ρυθμιστικές αρχές στην Ευρώπη. Ξέρω ότι οι συζητήσεις στη Γαλλία συνεχίζονται σε αυτή τη φάση. Δεν έχουν υπάρξει τελικές νομοθετικές προτάσεις. Ούτε από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακόμα. Τώρα, για τις κοινέ νομοθετικές ρυθμίσεις στον τομέα των πωλήσεων. Γνωρίζω την άποψη της ε, κυρία Γκέπχαρτ σε ό,τι αφορά το κοινό δίκαιο για τις πωλήσει. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Αυτό που ωστόσο είναι καινούριο είναι το ότι το Κοινοβούλιο έχει διενεργήσει δική του μελέτη αντικτύπου σε ό,τι αφορά το κοινό δίκαιο για τις πωλήσει. Και νομίζω ότι αυτή η μελέτη αντικτύπου είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ σημαντική. Γιατί τι σε τι καταλήγει, σε τι πορίσματα καταλήγει. Καταλήγει με σαφήνεια στο ότι η μελέτη αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εδώ πέρα αναφέρω και παραθέτω τι λέει η δική σας ε, μελέτη αντικτύπου είναι πάρα πολύ αξιόπιστη και πιστευτή. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφορές οι οποίες θα ληφθούν υπόψη ασφαλώ από το Κοινοβούλιο κατά τι διαπραγματεύσεις, αλλά σε γενικές γραμμές η μελέτη αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρείται από την ίδια τη μελέτη αντικτύπου του Κοινοβουλίου ω ως μια βάσιμη μελέτη αντικτύπου, Ω μια σωστή βάση και χάρηκα ιδιαίτερα όταν το διάβασα αυτό γιατί κάτι διαφορετικό, το αντίθετο μάλλον θα προκαλούσε προβλήματα. Προβλήματα για τις λεπτομέρειες υφίστανται. Και αυτό άλλωστε ε, πραγματεύονται στην παρούσα φάση η υπεύθυνη κατάρτιση της νομοθεσίας. Ε, νομίζω ότι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων είναι η καθήλυνα αρμόδια, προκειμένου να κρίνει το πώς η πρόταση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προκειμένου να αυξήσει τον ανταγωνισμό κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν τολμούν να βγουν έξω από τα σύνορα της χώρας τους σήμερα γιατί στην περίπτωση αυτή αναγκάζονται να εφαρμόσουν το δίκαιο της γειτονικής χώρας. Έτσι λοιπόν ο καταναλωτής θα έχει επιλογή ο καταναλωτής ο οποίος σήμερα σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει δικαίωμα καν να ψωνίσει εκτός του κράτους μέλους του, γιατί πολύ απλά δεν του προσφέρονται τα project αυτά και οι υπηρεσίες αυτές. Άρα θα ισχύσει και για τους ε, καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις. Θεωρώ ότι θα είναι ένα πλεονέκτημα και για τις δύο πλευρές και πραγματικά θέλω και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το πιστεύω αυτό, ότι θα επιλύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Κοιτάξτε, δεν ε, λέω ότι γνωρίζω και την απόλυτη αλήθεια σε ό,τι αφορά το οτιδήποτε. Θα κάνω μια πρόταση, πρόταση θα ακούσω και το Ευρωπαϊκό και το Συμβούλιο. Και για να το συνδέσω αυτό και με την ερώτηση που έθεσε η κυρία Ράπτη για το ADR. Το ADR και το ODR συμπεριλαμβάνονται στο κοινό δίκαιο για τις πωλήσει. Άρα υπάρχει καταρχάς η υποχρέωση να περάσουμε από αυτές τις μεθόδους προτού μπορεί κανείς να προσφύγει σε εθνικό δικαστήριο. Το οποίο και αυτό αποτελεί έναν ενδιαφέροντα τρόπο να προωθηθούν τα θέματα ADR και ODR. Το θέμα του collective redress, των συλλογικών αγωγών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποτέ δεν θεώρησε ότι ήταν αυτός σκοπός το θέμα των συλλογικών αγωγών. Πάντα το θεωρούσε ως ένα εργαλείο. Ένα εργαλείο για να επιτευχθούν οι στόχοι της πολιτικής της Ένωσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το σχετικό πρόγραμμα εργασίας του 2012 είχαν ως στόχο μία πρωτοβουλία, όχι όμως μία δράση προτεραιότητας και προκειμένου να συνάδει το έργο μας με αυτό το προπαρασκευαστικό έργο συνεχίζουμε να δουλεύουμε προς την κατεύθυνση αυτή και συνεργάζομαι στενά με τους συναδέλφους Αλμούνια, Μπός και μετά τη συνεργασία με τον Επιτροπό Ντάλι ανέλαβε τώρα ο Επιτροπός Μπός και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σχετικό ψήφισμα προς μια ευρωπαϊκή κοινή προσέγγιση για τις συλλογικές αγωγές λαμβάνεται στα σοβαρά υπόψη η πρόταση που θα καταθέσει δε ΔΕΗ Επιτροπή θα αποφύγει τα αρνητικά στοιχεία των άλλων μοντέλων δικαιοδοσίας. Να είστε σίγουροι και θα φροντίσει να προβλέψει εγγυήσει για τα μέρη και για τους μηχανισμούς που θα αποτρέψουν τέτοιες προβληματικές αγωγές. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Έχουμε μόλις ένα τέταρτο στην διάθεσή μα. Αν θέλετε λοιπόν να είστε πάρα πολύ σύντομοι στι ερωτήσει, να ακούσουμε τον επόμενο γύρο ερωτήσεων. Μάιερ, Σαλδεμόζα και. Μάιερ. Ο κύριο Μάιερ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, η έκθεση αξιολόγηση και η διαπίωση της νομικής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι επαρκή για μένα για να θεωρήσω ότι έχει λυθεί το θέμα του αν θέλουμε να προχωρήσουμε ή όχι. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μια μεγάλη αγορά, μια μεγάλη παραγωγή, παράγουμε το 1 τέταρτο της παγκοσμίας παραγωγής. Και εκ των έξω μας θεωρούν σαν μια τεράστια εμπορική ενότητα. Βλέπουμε όμως ως Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς ότι δεν λειτουργεί ακόμα πλήρως και όπως θα έπρεπε η εσωτερική αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ είμαι τώρα συνεισηγητής για τα δικαιώματα των αγοραστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για το δίκαιο των αγορών και εδώ έχουμε μεγάλα εμπόδια τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι φυσικά το μοναδικό εμπόδιο, αλλά είναι ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια τα οποία δεν επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Ενία Αγορά να λειτουργήσει και την κατακαιρματίζει σε 27 διαφορετικά εθνικά δικαιακά σε δικαιακούς χώρους. Το ερώτημα είναι λοιπόν πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα λειτουργήσει καλύτερα η εσωτερική αγορά για το όφελος του καταναλωτή. Ε, εγώ πιστεύω ότι ναι πρέπει να το πετύχουμε αυτό γιατί ο καθένας από τους 500 τα 500 εκατομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένας δυνητικός ε, αγοραστής και δυνητικός καταναλωτής. Επομένως, δεν μας ενδιαφέρει μονάχα το γεγονός ότι έχουμε μια εμπορική ικανότητα, πρέπει να έχουμε και την προστασία των 500 εκατομμυρίων καταναλωτών από το επιγραμμικό εμπόριο ο καθένας από εμά μπορεί να διαπιστώσει ότι ποτέ δεν υπάρχει μια εταιρεία που να πουλάει σε παραπάνω από 10 χρόνια. Ποτέ στις 27 χώρες. Δεν είναι μόνο τα γλωσσικά προβλήματα τα οποία εμποδίζουν αυτό. Σε 10 χώρες που πουλούν οι περισσότερες εταιρείες ήδη πρέπει να λειτουργούν σε 8 γλώσσε περισσότερες φορές. Επομένως δεν είναι η γλώσσα η οποία αποτελεί το πραγματικό πρόσκομα για να υπάρξει δυνατότητα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως αυτό το δίκαιο ε, για τις αγορές ε, δίνει περισσότερη έμφαση στο, στα δικαιώματα των καταναλωτών αλλά όχι επαρκή προσέγγιση για τα ζητήματα των ε, εμπόρων και τις, ε, τα εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζουμε. Εμείς θεωρώ ότι πρέπει να βασιστούμε σε δύο βασικές έννοιες, τον πολιτή και τον καταναλωτή και να εστιάσουμε εκεί. Αν λοιπόν δημιουργήσουμε ένα επαρκές πλαίσιο για τις πωλήσει αυτές και μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη και τις ανάγκες των καταναλωτών, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Δεύτερον, τα θέματα των, του, το διαδικαστικού κόστους έχει καταρχήν επιληθεί, αλλά εδώ χρειάζεται να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή της Κομισιόν. έχουμε τη δυνατότητα της εξοδικαστικής επίλυσης ε, διαφορών. Αλλά εκεί υπάρχουν ε, ακόμα δυσκολίες. Και έχουμε και τις διαδικασίες για την εφαρμογή αποφάσεων όταν υπάρξει πραγματική διαμάχη και δεν υπάρξει συνενετική λύση, αλλά όλα αυτά επισύρουν ένα κόστος διαδικαστικό το οποίο δεν είναι γνωστό. Δεν το γνωρίζουν ακόμα και οι οι δικηγόροι σε όλες τις περιπτώσεις. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να ξέρει κανείς, γιατί εγώ δεν μπορώ να πάω σε ένα δικαστήριο και να πάρω λεπτομέρειες για το πόσο θα κοστίσει αυτή η διαδικασία επίλυσης μιας διαφοράς. Εντάξει, μιλάμε πολύ για τα θέματα τα οποία επιλύουμε με τις ρυθμίσεις αυτές, αλλά οι απλοί πολίτες και οι απλοί έμποροι θέλουν να ξέρουν τι, σε τι θα τους ωφελήσει όλη αυτή η διαδικασία. Γι' αυτό είναι το δεύτερο ερώτημα το οποίο θέλω να θέσω. Θεωρεί η Κομισιόν ότι θα μπορέσει σύντομα και με ενεργητικό τρόπο να ξεκινήσει μια εκστατεία πληροφόρηση για τα θέματα αυτά, για τις επιλύσεις διαφορών κτλ. Ευχαριστώ κύριο Σαντεμόσερ. Σας ευχαριστώ. Περισσότερο ένα σχόλιο θα να κάνω παρά να θέσω ένα ερώτημα. Συμφωνώ μαζί σας ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτες και οι καταναλωτές έχουν εμπιστοσύνη στην εσωτερική αγορά, αλλιώς δεν θα την χρησιμοποιήσαμε. Είδαμε με το αλογίσιο κρέας ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο και ζωτικό να πιστεύουν αυτά που τους λένε οι πολιτές και οι εταιρείε. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να πούν οι Κομισιόν και τα κράτη-μέλη στους καταναλωτές ποια είναι τα δικαιώματα που έχουν ήδη σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι μια κεντρική εκστρατεία από την Κομισιόν δεν θα ήταν ίσως ο μόνος τρόπος πληροφόρησης των καταναλωτών. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος πληροφόρησης των καταναλωτών είναι τα ισχυρά συμβούλια καταναλωτών σε εθνικό επίπεδο, γιατί αυτή είναι πολύ πιο κοντά στον απλό καταναλωτή. Επίσης και τα κοινωνικά μέσα διαδικτύωσης μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο για να μεταφέρουν στους καταναλωτές τις ειδήσει αυτές. Εγώ στο Facebook έβαλα στη σελίδα μου για την απόφαση της ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα των Επιβατών. Είναι ένα τρόπο με τον οποίο μπορούν να γνωρίζουν οι καταναλωτέ ποια είναι τα δικαιώματά του και να τα χρησιμοποιούν περισσότερο. Πρέπει, εγώ πιστεύω όμω, να καταστεί σαφέ πού βρίσκεται η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και εδώ η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο μπορούν να δώσουν ο ένας τον άλλο αμοιβαία αρρωγή, γιατί είναι κεφαλαιότητε για τον Ευρωπαίο πολίτη να καταλαβαίνει από πού προέρχεται η ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Σας ευχαριστώ πάντως για όλα αυτά που μας λέτε και τις προσπαθίες σας. Ευχαριστούμε κυρία Βάιλερ. Ναι. Και εγώ από πλευρά μου επιβεβαιώνω ότι τα πράγματα είναι όπως είπε η Κρίστελ. Οι καταναλωτέ θα ήθελαν να υπάρχουν σαφείς κανόνες. Να μην είναι πάρα πολύ περίπλοκα τα πράγματα. Στη δική μου χώρα, στη Γερμανία, ε, που τα πράγματα ε, ήταν τόσο σαφέστατα στην αρχή κατά τη σηματοδότηση αυτή με τα χρώματα, Τώρα ο κόσμος έχει αλλάξει νοοτροπία. Ιδιαίτερα μετά το σκάνδαλο με το αλλαγή κρέα, ε, θεωρώ ότι καλό θα ήταν να αλλάξει κάτι. Όπως και να έχει. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργαστεί το θέμα αυτό. Να έρθω σε θέματα χρονοδιαγράμματος. Δεν έχουμε χρόνο, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πλέον πολύ χρόνο να καταρτήσει νομοθεσία η οποία θα εφαρμοστεί μέχρι τα τέλη της θητείας. Αν θέλουμε μέχρι τα τέλη της θητείας να περάσει κάτι ουσιαστικό, θα πρέπει να το έχουμε δρομολογήσει μέχρι το Πάσχα. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ, όπως είπε και η συνάδελφος Ράπτη, τα θέματα collective redress συλλογικών αγωγών. Άκουσα πόσο ήπια απαντήσατε ότι δεν είναι ο σκοπός αυτός, ότι είναι ένα εργαλείο κτλ. Και ότι θα πρέπει να μην γίνουν καταχρήσεις. Συμφωνούμε, συμφωνούμε όλοι εδώ πέρα στο Κοινοβούλιο. Δεν θέλουμε το αμερικανικό μοντέλο, θέλουμε ένα ευφυές ευρωπαϊκό μοντέλο. Αλλά θέλουμε να υπάρχει ένα μοντέλο. Και στην αρχή της θητείας τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μας ε, έλεγαν ότι υπάρχει διάθεση να κάνουμε κάτι. Δεν ξέρω αν έκανα, αν άκουσα σωστά. Τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα χρονοδιάγραμμα για ευρωπαϊκή νομοθεσία, όχι για αμερικανικό μοντέλο, προκειμένου να μπορέσουμε να το ψηφίσουμε και στην Επιτροπή μέχρι τα τέλη του χρόνου και στην Ολομέλεια μέχρι ε, το, την Άνοιξη. Γιατί μετά θα έχει τελειώσει ουσιαστικά. Γιατί ιδάλω θα έχουμε χάσει, θα έχουμε καθυστερήσει πέντε χρόνια. Commissioner. The Για uh, ε, την πρώτη ερώτηση για την ρύθμιση την νομική για τις πωλήσει. Χαίρομαι γιατί το Κοινοβούλιο στα πλαίσια των επιτροπών του εξετάζει και βρίσκει ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ένα χρήσιμο μέσο στην ουσία θα έπρεπε να αναφερθούμε σε αυτή τη ρύθμιση όχι απλά σαν μια ρύθμιση αλλά σαν δίκαιο ειδικό για, που εφαρμόζεται στην περίπτωση των πολίσεων και έτσι και οι πολίτες θα ενημερωθούν καλύτερα για την ύπαρξη αυτών των μορφών δικαίου. Οι πολίτες θα κατανοήσουν σύντομα εφόσον συμφωνήσει βέβαια το Συμβούλιο με το Κοινοβούλιο οι πολίτες λοιπόν πάρα πολύ σύντομα θα κατανοήσουν ότι τα αγαθά τα οποία δεν μπορούσαν στο παρελθόν να αγοράσουν online, τώρα ε, θα μπορέσουν να το κάνουν εφόσον ε, το επιθυμούν. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ένα σημαντικό μήνυμα και έχετε απόλυτος δίκιο λέγοντας ότι γίνονται σε αυτή τη φάση κάποιες, ρυθμίσεις, τις, κάποιες αλλαγές στις νομοθετικές ρυθμίσεις. Έχουμε όμως μια σωστή, όπως λέμε, εργαλειοθήκη, ένα σωστό toolbox. Έχουμε τα μέσα. Όταν γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για τα εδάφη τους, έτσι ώστε να δημοσιοποιήσουν τα διαθέσιμα μέσα και τις ισχύουσες νομοθετικές τους ρυθμίσεις. Δυστυχώς όμως όταν συζητώ με τους καταναλωτές δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά τα κράτη-μέλη ως προς αυτό. Δεν λέω ότι δεν κάνουν προσπάθειες. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι μια μεγάλη εκστρατεία πληροφόρησης η οποία θα επεξηγεί τα δικαιώματα των καταναλωτών, των πολιτών, θα ήταν πολύ σημαντική. Θα ήταν πολύ σημαντική και για το Κοινοβούλιο, γιατί αυτό θα ήταν ένα καλό μέσο ε, και για την προεκλογική εκστρατεία. Θα μπορέσετε να δείξετε το τι κάνει το Κοινοβούλιο για να ενισχύσει τους πολίτες ως καταναλωτές στα κράτη-μέλη τους και εκτός αυτών. Ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστές αυτές οι νομικές ρυθμίσεις είναι επίσης γιατί οι ίδιοι οι δικηγόροι ο κόσμος της δικαιοσύνης δεν γνωρίζουν απόλυτα την ύπαρξη αυτών των νομικών ρυθμίσεων. Και γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει την κατάρτιση όχι μόνο δικηγόρων, αλλά και εκπροσώπων του δικαστικού. Για το σύνολο των ευρωπαϊκών δικαϊκών ρυθμίσεων. Γιατί οι εθνικοί εμπειρογνώμονες είναι εμπειρογνώμονες στο εθνικό δίκαιο συνήθως και δεν γνωρίζουν το τι ισχύει στις υπόλοιπες χώρες. Και γι' αυτό ακριβώς και έχουμε δημιουργήσει και την θύρα στο διαδίκτυο e-justice, έτσι ώστε να μπορούν οι δικαστές να βλέπουν τι ισχύει στις γειτονικέ χώρες, γιατί πολλές φορές καλούνται τελικά να εφαρμόσουν νομοθετικές ρυθμίσεις διαφορετικές από τις εθνικές τους. Και γι' αυτό ακριβώς αυτά τα δίκτυα που έχουμε δημιουργήσει είναι σημαντικά. όχι ότι ο δικαστής να γνωρίζει ε, το τι ακριβώς συμβαίνει και το τι ακριβώς ισχύει στη γειτονική χώρα, αλλά να μπορεί να γνωρίζει και να έλθει σε επαφή με κάποιον στη γειτονική χώρα που το κάνει αυτό, που μπορεί να τον ενημερώσει. Έτσι λοιπόν θέλουμε να έχουμε και ισχυρές οργανώσεις καταναλωτών. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα μέλος, το Λουξεμβούργο, που η οργάνωση των καταναλωτών είναι ισχυροτάτη και σχεδόν όλος ο κόσμος την γνωρίζει. Ε, δυστυχώς αυτό δεν ισχύει σε όλες τις χώρες. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να γνωστοποιήσουμε καλύτερα τη δράση μας. Υπάρχει και αυτή η νέα θύρα στο διαδίκτυο που λέγεται U Europe, την οποία εγκατέστησα από κοινού με τον Μισελ Μπαρνιέ. Πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια των δύο επιτρόπων ο ένας ασχολείται με την εσωτερική αγορά και ο άλλος ασχολείται με τους πολίτες καταναλωτές. Έχουν οι πολίτες λοιπόν μία θύρα στο διαδίκτυο, μπορούν να καταθέσουν τις ερωτήσεις τους, ακόμα και πολύ περίπλοκες ερωτήσεις, οι οποίες θα παραπευθούν στις πλέον αρμόδιες των υπηρεσιών, αλλά είναι σαφές ότι οι πολίτες θα πάρουν μία απάντηση δεδομένη από το σύστημα αυτό. Έχει μεγάλη σημασία αυτό και είναι διαθέσιμο τώρα πλέον σε όλες τις γλώσσες. Προσπαθήσαμε λοιπόν και ξεκινήσαμε και μια εκστρατεία πληροφόρησης στις διάφορες χώρες μέλη για να πούμε το τι υπάρχει και το τι είναι διαθέσιμο σήμερα. Παρ' όλα αυτά όταν πηγαίνω στις χώρες και ερωτώ τους πολίτες για το τι γνωρίζουν γύρω από αυτό δυστυχώς το επίπεδο γνώσεων είναι πολύ χαμηλό και πρέπει σαφώς να καταστούμε αποτελεσματικότεροι μέχρι το τέλος του χρόνου και τις αρχές του επομένου, έτσι ώστε πριν ξεκινήσετε την προεκλογική σας εκστρατεία να έχετε προχωρήσει σε συντονισμένες μορφές ε, δημοσιοποίησης. Χαίρομαι που συνεργάζομαι με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το θέμα εδώ δεν είναι νομικών αντιπαραθέσεων. Το θέμα εδώ είναι να προωθήσουμε την Ευρώπη και να συνεργαστούμε. Τώρα να έρθω στην ερώτηση της συλλογική προσφυγής. Ο Χωακίν Αλμούνια, ο συνάδελφος, θα ασχοληθούμε, θα προωθήσουμε μάλλον, θα πάρουμε μια πρωτοβουλία εν πάση περιπτώσει και θα δώσουμε μια συνέχεια στις διαβουλεύσεις που έχουν ξεκινήσει πριν από το τέλος της περίοδου. Όπως είπα, έχουμε σημειώσει προσεκτικά το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις συλλογικές προσφυγές και θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε και τις δικές σας προτάσεις στην δική μας και θα σας την καταφέσουμε. Καλώς, τώρα πλέον δεν έχουμε χρόνο. Θα ήθελα να έχουμε χρόνο για να μιλήσουμε και με την κυρία Γένσεν μετά που είναι το επόμενο θέμα μας και ξέρω ότι δεν έχει πολύ χρόνο. Αλλά για τον κύριο Ροσφόρ και τον κύριο Σβάμπ. Παρακαλώ ένα λεπτό ο καθένας, όχι παραπάνω. Ο κύριος Ροσφόρ πρώτος. Πάρα πολύ γρήγορα κύριε Πρόεδρο. Σας ευχαριστώ για τη σαφήνεια των λόγων σας κυρία Επίτροπε. Καταδεικνύεται πόσο είναι προσφυλές σε εσά και πόσο είναι σημαντικό σε εσά να εξασφαλιστεί η προστασία του καταναλωτή. Είναι το κέντρο της φιλοσοφίας σας. Εγώ θέλω να εστιάσω τώρα στη μεταγραφή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών. Επί της ουσίας, στη δική μου χώρα, στη Γαλλία, αυτή η μεταγραφή είναι εν εξελίξη, θα υπάρξει ένα νομοσχέδιο σχετικά. όπω πάντα ο Γάλλος υπουργό θα πει ότι είναι τα νέα δικαιώματα που δίνει η Γαλλία στου Γάλλου καταναλωτέ. τα έχουμε συνηθίσει αυτά, δεν μα πειράζει. Αυτό όμως το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι υπάρχουν δύο είδη νέων δικαιωμάτων. Υπάρχουν τα νομικά δικαιώματα, υπάρχει καλύτερη προστασία σε νομικό επίπεδο, αλλά και οικονομικά δικαιώματα. Δηλαδή ο καταναλωτής μέσω αυτής της εναρμόνιση θα μπορεί να αγοράζει από ιστοσελίδε που είναι έξω από τη χώρα του και σε άλλου χώρου, λοιπόν από του εθνικού χώρου. Εγώ πιστεύω ότι οι περισσότερες κυβερνήσεις δεν θα δώσουν αυτή τη δυνατότητα. Θα πούν βεβαίως υπάρχουν νέα δικαιώματα, όλα αυτά τα κάνει η Ευρώπη ή τα, κάνει, τα κάνουμε εμείς καλύτερα, αλλά δεν νομίζω ότι θα κάνουν όλα αυτά που είναι απαραίτητα ώστε να μπορούν οι πολίτες να βγαίνουν από τον εθνικό χώρο και εθνικό διαδικτυακό χώρο γιατί για μια μεγάλη χώρα όπως η Γαλλία, το ίδιο ισχύει για τη Γερμανία και την Αγγλία, ίσως κύριε Πρόεδρε το γνωρίζω, Οι χώρες αυτές είναι τόσο μεγάλες που οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν θέλουν να υπάρξει μια τέτοια διευκόλυνση. Θέλουν να υπάρξει ο εθνικό κατακαιρματισμό. Πολλέ μικρομεσαίε επιχειρήσει όμω θα μπορούσαν να ευνοηθούν αν είχαν τη δυνατότητα να πολλούν σε καταναλωτέ εκτό τη της χώρα του, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ζητώ λοιπόν να υπάρξει αυτή η προσπάθεια καλύτερη επικοινωνία, αλλά αυτή η προσπάθεια επικοινωνία δεν πρέπει να αφορά μοναχα την πρόσβαση στα νέα δικαιώματα, γιατί σε πολλέ χώρε αυτό έχει ήδη επιτευχθεί, αλλά και την πρόσβαση, αν θέλετε να το πω έτσι, στα οικονομικά δικαιώματα. Δηλαδή το, να μπορεί ο καταναλωτή να έχει πρόσβαση σε άλλου χώρου όπου μπορεί να κάνει αγορέ. Σα ευχαριστώ, λέει ο για αυτό το διαπεραστικό ερώτημα. Η γαλλική κυβέρνηση βέβαια δεν είναι η μόνη η οποία λέει στους καταναλωτές ότι αυτή προσφέρει τα δικαιώματα στους καταναλωτές που τελικά απορρέουν από τη συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Φάμπος εισηγητής. Ε, ε ευχαριστώ. Μετά από αυτά που ελέγχθησαν δεν χρειάζεται να μακρηγορήσω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί η νομοθεσία αυτή στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε είναι κάτι αντίστοιχο με την οδηγία για τις ε, αθέμητες πρακτικές σε χρηματοπιστωτικά θέματα. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσετε κύριε Επίτροπε ότι θα γίνει αυτό το θέμα με σωστό τρόπο η μεταγραφή και ξέρω ότι το παρακολουθείτε ήδη. Δεύτερον, εγώ μίλησα με ένα Ισπανό ο οποίος εκπροσωπεί μια μικρομεσαία επιχειρήση και λέει ότι δεν μπορούν να πωλήσουν προϊόντα τα οποία είναι φθαρτά σε γειτονικέ χώρες, νοπά ε, τρόφιμα παραδείγματο χάρη και είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάρει κάποια απο, απάντηση από εσά γιατί θα πρέπει να ισχύει ε, και για τα πορτοκάλια και για τα λεμόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση όπω λέει ο κ. Το τελευταίο σημείο που θέλω να θίξω είναι ότι για τα κέντρα των καταναλωτών στην Ευρώπη είναι πολύ διαφορετική η προσέγγιση στην ε, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τρόπο με τον οποίο κατατάσσουν τα δικαιώματα που έχουν να κάνουν με την εξασφάλιση του ανταγωνισμού. Και επομένως θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση σε αυτά τα θέματα για να μην υπάρξει πρόβλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Βίβιαν, θέλετε να απαντήσετε. Για το τελευταίο ερώτημα του κυρίου Σβάμπ υπογραμμίσατε τα θέματα αυτά, αλλά πρέπει να τα εξετάσω. Μου προκαλεί έκπληξη. Μου προκαλεί έκπληξη. Αλλά θα πρέπει να το εξετάσω, γιατί εγώ αυτό που είδα και βλέπω με την προσωπική μου εμπειρία και ως πολιτικός και σε εθνικό επίπεδο είναι το εξής. Οι οργανώσεις αυτές όταν παίζουν σωστά το ρόλο τους είναι πάρα πολύ σημαντικές γιατί ουσιαστικά κάποια προβλήματα δεν τα αφήνουν να φτάσουν στο δικαστήριο γιατί παίζουν το ρόλο του μεσάζοντα. Αποτελούν ένα σημαντικό φορέα μεταξύ του πολιτή και του αγοραστή για την εφαρμογή της οδηγίας. Φυσικά, η εφαρμογή όλων των οδηγιών αποτελεί θέμα υψής της σημασίας. Δεν μπορώ τώρα να σας πω στις πιο πολλές περιπτώσεις τα κράτη-μέλη σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους και δεν εμφανίζεται ποτέ η Ευρώπη. Και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί σε κάποιες περιπτώσεις διαβάζω στον τύπο ότι ένα, ένας καινούριος ε, νόμος ε, καταρτίστηκε και ε, σκέφτομαι ότι κάπου τον έχω δει, κάπου τον έχω ακούσει και πρόκειται για όταν το κοιτάω καλύτερα, διαπιστώνω ότι πρόκειται για μια εφαρμογή οδηγίας, αλλά αυτό που δεν άδεν αναφέρεται και αυτό ισχύει σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις. Δεν μου προκαλεί εντύπωση, έτσι έχει ζωή, τι να κάνουμε. Προσπαθούμε όμως να ενημερώνουμε όσο πιο πολύ γίνεται και γι' αυτό λοιπόν θα είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η κοινή ενημερωτική εκστρατεία και αυτό που είπατε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για την δυνατότητα να κάνουν πωλήσει σε διασυνοριακό επίπεδο. Αυτό ελπίζω, ελπίζω, αν συμφωνήσουν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ελπίζω να επιληθεί στο δίκαιο για τις πωλήσει γιατί θα επιτρέψει κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κάνουν συναλλαγές διασυνοριακά χωρίς το δυσανάλογο κόστος της προσαρμογής στο δίκαιο της γειτονικής χώρας και τελικά το αποτέλεσμα να είναι ότι ο κόσμος δεν μπορεί να αγοράσει προϊόντα σε διασυνοριακό επίπεδο. Αυτό προφανώς ε, διαφέρει πολύ στις μεγάλες χώρες από ό,τι στις μικρές, γιατί στις μεγάλες χώρες υπάρχει μία μεγάλη ενιαία αγορά και ως πολιτής προσπαθεί κανείς να προσαρμοστεί στο δίκαιο μιας μεγάλης χώρας. Αυτό δεν συμβαίνει προφανώς ε, για τις μικρές χώρες, άρα είναι πολύ διαφορετικός ο βαθμός της εφαρμογής της νομοθεσίας. Και αυτό αφορά ασφαλώς και τα δικαιώματα του καταναλωτή, γιατί κάποιοι καταναλωτές σε μικρές χώρες πολύ απλά δεν μπορούν να αγοράσουν γιατί δεν τους πουλάνε οι πολιτές. Θα θέλω λοιπόν, θα ήθελα να υπάρχει ίσο επίπεδο για όλες τις χώρες και παρεπιπτόντως θεωρώ ότι ο κόσμος του διαδικτύου θα αναπτυχθεί πολύ περισσότερο. Σήμερα 6% των πολιτών αγοράζουν διασυνοριακά μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο είναι παράλογο, αλλά και πάλι συνδέεται με τα προβλήματα αυτά. Ελπίζω. Αύριο, όταν θα έχουν μεγαλώσει οι σημερινοί πολίτες που έχουν μεγαλώσει με το ίντερνετ, αυτό να μην αποτελεί πλέον εμπόδιο και να μπορούν να κάνουν συναλλαγές οπουδήποτε το επιθυμούν στην Ευρώπη. Συμφωνώ απόλυτα με το ότι η εφαρμογή του νόμου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά Πρόκειται για κάτι το οποίο είναι πολύ κοστοβόρο σε ό,τι αφορά το προσωπικό. Ως Επίτροπος εξέτασα κάποιες από τις οδηγίες ε, που έχουν εφαρμοστεί εδώ και πολύ καιρό και διαπιστώνω ότι τα πιο πολλά κράτη-μέλη δεν τις έχουν εφαρμόσει όπως θα έπρεπε. Ε, στην περίπτωση αυτή λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουν ατέρμονες συζητήσεις οι οποίες παίρνουν και χρόνια προτού τελικά προσαχθεί και το τελευταίο κράτος μέλος που δεν έχει εφαρμόσει την νομοθεσία και αυτό καταλαβαίνετε τι κάνει σε ό,τι αφορά την δημοτικότητά μου ως επίτροπο στα κράτη-μέλη. Είμαι πάρα πολύ... Έχω μεγάλα προβλήματα δημοτικότητας γιατί παρακολουθώ τέτοια στοιχεία τα οποία αποτελούν όμως τη βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχω πραγματικά προσάγει κράτη-μέλη και κύριε ΣΒΑΠ για το θέμα με τα πορτοκάλια που αναφέρατε. Λίαν συντόμπος, θα σας αποστείλω μία απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Όπως πάντα, είναι πάρα πολύ σαφή τα σχόλιά σας και πολύ καλή η γνώση σας ε, για όλους τους τα θέματα και ο ενθουσιασμός σας είναι πασιφανής. Δεν έχετε πρόβλημα δημοτικότητας ε, σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη. Ε, εν πάση περιπτώσει, σε εμά, στο Κοινοβούλιο είστε πάρα πολύ δημοφιλεί. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μα χαρά που σα είχαμε μαζί σήμερα το απόγευμα και θα λάβετε ασφαλώ πάρα, πάρα πολλά σχόλια και τα κράτη-μέλη. Good. Um να προχωρήσουμε και πολύ λυπάμαι που δεν μπόρεσα να συνοδεύσω έξω την κυρία Ρέντιν γιατί είμαστε στη μεγάλη αίθουσα, στην μεγάλη αίθουσα και ξέρω ότι η κυρία Γέντσεν αντιμετωπίζει και αυτή η χρονική πίεση. Να ξεκινήσει λοιπόν η συζήτηση για τον προπολογισμό του 2014 Γενική συγγήτρια είναι η κυρία Αν Γένσεν, όπως σας είπα θα κάνει μια εισαγωγή. Νομίζω ότι δεν έχουμε λάβει υποψηφίους από τις ομάδες ακόμα. Να ρωτήσω αν θέλει να πάρει το λόγο ο κύριος Σφάπ. Να δούμε ποιον έχουν ορίσει οι ομάδες και ποιον, ποιον θέλουν, σε ποιον θέλουν να δώσουν χρονομιλία. Αλλά να κάνει κάποια εισαγωγικά σχόλια καταρχάς η κυρία Αν Well, thank you very uh, Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να θέσω το πλαίσιο για τον προϋπολογισμό του 2014. Το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι δεν έχουμε ένα πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ακόμη. Δεν έχουμε την ομοθετική βάση για τον προϋπολογισμό του επομένου έτους, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να περάσουμε σε ένα ψήφισμα σε σχέση με το τι θα περιμένουμε από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και έτσι θα έχουμε και τη δυνατότητα να ορίσουμε το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Ιρλανδική πλέον Προεδρία. πέρα από τις διαπραγματεύσεις για τα συγκεκριμένα ποσά και για το πώς θα προχωρήσουμε σε αιτήσια δημοσιονομική βάση, έχουμε πάρα πολλά θέματα πάνω στα οποία θα κληθούμε να πάρουμε αποφάσεις. Η Ιρλανδική Προεδρία είπε ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις παρά μόνο μετά την 22 Απριλίου. Οπότε θα χρειαστεί να φτάσουμε Ιούνιο ή Ιούλιο πριν τελικά υπάρξει κάποια συμφωνία για το πολιετές δημοσιονομικό. Τώρα η Επιτροπή θα κάνει μία πρόταση τον Μάιο, μέσα Μαΐου, το είπαν αυτό, το ανακοίνωσαν. Στην ανακοίνωσή τους θα βασιστούν στη δική τους πρόταση για το πολιετές δημοσιονομικό, την οποία γνωρίζετε τουλάχιστον στους τομείς που αφορούν την Επιτροπή σας. έχετε ασχοληθεί με τα θέματα που σας ενδιαφέρουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σημείωσε ότι έχει υπάρξει, ε, λαμβάνει υπόψη μάλλον, τη συνάντηση των ε, ηγετών των κρατών μελών γύρω από τα θέματα του προϋπολογισμού και αυτά θα ληφθούν υπόψη στις προτάσεις της για τον προϋπολογισμό του 2014. Όταν ανακοινώσει αυτά η Επιτροπή θα ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Κοιτάξτε, ε, θα πρέπει να πω ότι από τις 19 Μαρτίου θα υπάρξει ένας ανεπίσημος τριμερής διάλογος ανάμεσα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Το θέμα θα είναι η μεθοδολογία των διαπραγματεύσεων για τον ετήσιο προϋπολογισμό. Τα τελευταία τρία χρόνια, στα πλαίσια λοιπόν της ρύθμισης που προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας, Είδαμε ότι το Συμβούλιο ξεκίναγε ε, τις διαπραγματεύσεις την τελευταία μέρα που μπορούσε να το κάνει, ή τα μεσάνυχτα της 21ης Απριλίου κάθε φορά. Λοιπόν, δεν υπάρχει μια τέτοια συμφωνία κατελάχιστον σε αυτή τη φάση και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε προτάσεις για καλύτερους τρόπους διαπραγμάτευσης και ίσως λοιπόν να μπορέσουμε να έχουμε μια συζήτηση για τα θέματα αυτά στις 19 Μαρτίου. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν, σαν εισηγήτρια εγώ, να είμαι σε στενή επαφή και σε διάλογο με τις διάφορες επιτροπές του Κοινοβουλίου, έτσι ώστε να γνωρίζω σωστά τις προτεραιότητές σας. Έχουμε ήδη κάποιες κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες έχουν γίνει αντικείμενο ψηφοφοριών στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και θα φτάσουν στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα. Σε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές το Κοινοβούλιο ζητά να υπάρξει μια λύση για τις πληρωμές. Ακούσαμε κάποια σχόλια για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων για το πολιετές δημοσιονομικό και είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη στροφή στην ανάπτυξη και στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Μπορούμε να γίνουμε πιο, θα έλεγα, συγκεκριμένοι ε, για τα θέματα τα οποία θα έρθουν προς συζήτηση αργότερα. Το Συμβούλιο έχει και αυτό προχωρήσει σε ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές λέγουν ότι είμαστε σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση και ότι δεν θα πρέπει να δαπανίσουμε πάρα πολλά χρήματα, αλλά από την άλλη έτσι και αλλιώς αναγνωρίζει το ότι απαιτείται ανάπτυξη. Θα ήθελα λοιπόν εγώ να ακούσω τις δικές σας ιδέες και τις δικές σας αντιδράσεις. Ξέρω ότι εσείς εμένετε στα προγράμματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επίσης και για τα διευρωπαϊκά δίκτυα που αφορούν τις τηλεπικοινωνίες και την προστασία των καταναλωτών. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ και στη μεγάλη σημασία που έχουν τα προπαρασκευαστικά προγράμματα και δράσεις. Απαιτείται να γνωρίζουμε τις ιδέες σας, να γνωρίζω εγώ σαν ησυχήτρια τις ιδέες σας, όταν κάποια στιγμή ξεκινήσουμε τις συζητήσεις για τις προπαρασκευαστικές δράσεις το μήνα Μάιο. Ο κύριος Σβάμπ μου ανέφερε κάποιες λεπτομέρειες. Ξέρω ότι τα ποσά τα οποία σας ενδιαφέρουν δεν είναι πάρα πολύ υψηλά, αλλά βλέπουμε ότι μερικές φορές τα καλύτερα επιτεύγματα σημειώνονται στις μικρότερες γραμμές. Γι' αυτό λοιπόν τα σχόλιά σας θα μου είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Δεν ξέρω η χρήση της λέξης "chip" στα αγγλικά, ευθυμής. Κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε τόσο απαιτητικοί σε επίπεδο πόρων, αλλά αναμένουμε πάρα πολλά σε επίπεδο απόδοσης. Λοιπόν, ο κύριος Σβάμπ αυτό διορίστηκε από πλευράς Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σχολιαστής για τον προϋπολογισμό του 2014 και μετά και οι υπόλοιπε πολιτικές ομάδες, δεν ξέρω αν και αυτές θέλουν να αυτοπροσδιοριστούν οι συγητές, θα έχουν το λόγο. Λοιπόν, κύριο Βαμ πρώτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο διευκρινήσει να κάνω. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τις τιμές, τη λέξη «preiswert» στα γερμανικά, γιατί σίγουρα δεν είμαστε ευθυνοί εδώ πέρα στην Επιτροπή ε, προστασίας του καταναλωτή. Άρα, κυρία Γέντσεν, να διευκρινίσω αυτή την παρανόηση. Κατά δεύτερον, εγώ ούτε αυτοδιορίστηκα, ούτε με διόρισε κανένας άλλος εισηγητή. Αλλά είμαι μεσάζοντας, αν θέλετε, γιατί από, για οργανωτικούς λόγους ε, το ΕΛΚ δεν έχει διορίσει κάποιον υπεύθυνο εισηγητή, αλλά θα ήθελα τρία πράγματα να πω ε, επί της ουσίας ε, από πλευράς του ΕΛΚ σε ό,τι αφορά την, ε, το ψήφισμα της κυρίας Γένσεν. Η πρόταση που έχουμε μπροστά μας είναι όντως γενικόλογη και όπως είπε η κυρία Γένσεν, οι διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Γι' αυτό λοιπόν, ό,τι και να πούμε, είμαστε κάπως πρόοροι. Κατά δεύτερον, καλωσορίζουμε το γενικό, γενικά το γεγονός ότι υπάρχει το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και ότι υπάρχει δυνατότητα ε, θετικής ε, επιρροής του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στον παραγράφο 22 ιδιαίτερα, όπου προσπαθούμε να παίξουμε ένα ρόλο καταρρυντικό σε ό,τι αφορά τον ε, Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό για την ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και σημαντικό είναι λοιπόν το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο εδώ. Τρίτον, Πρόεδρε, φυσικά υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες οι οποίες αναφέρθηκαν και από την κυρία Γέντσεν άλλωστε. Εμείς θέλουμε προπαντός να ελεγχθεί το εξή. Όπως και τα προηγούμενα έτη και με τους προηγούμενους ε, προϋπολογισμούς, ε, το θέμα της κατανομής των πόρων και μεταξύ άλλων θέματα εθνικών εποπτικών αρχών. Θέλουμε το Solvit να συνεργαστεί με θέματα και εργαλεία ιστορικής αγοράς και θέλουμε επίσης τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτή να διατηρηθούν στο επίπεδο που βρίσκονται γιατί αυτό που είναι σημαντικό στην τελική ανάλυση είναι τα νομοθετήματα που βρίσκονται τώρα στο επίπεδο του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την ενία στην ενιαία αγορά κτλ. Αλλά και θέματα εφαρμογής, όπως το κόσμο. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτά τα ζητήματα είναι θέματα προτεραιότητας και θα θέλαμε να τα λάβει υπόψη η συγγήτρια και παρακαλούμε ασφαλώς και την ε, Επιτροπή και τα μέλη της Επιτροπής να υποστηρίξουν τις προτεραιότητες μας αυτές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μάλιστα, πολύ ωραία, λέει ο Πρόεδρος. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για το πλαίσιο. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς άλλος από κάποια άλλη ομάδα να πάρει το λόγο. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει οποιαδήποτε διαφωνία για τη γενικότερη κατεύθυνση που αναφέρεται. Το θέμα αυτό της προστιθέμενης αξίας είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα σε τομείς όπως τα προγράμματα και η ενημέρωση των ε, καταναλωτών, θέματα που συζητήσαμε και με την κυρία Ρέντινγκ, ε, το ευρωπαϊκό, ο ευρωπαϊκός κόμβος στο διαδίκτυο. Όλα αυτά θα είναι πάρα πολύ σημαντικά αν θέλουμε να υπάρχει απόδοση της νομοθεσίας μας. Να υπάρχει απόδοση της επένδυσης Κυρία Γένσεν, θέλετε να πάρετε το λόγο ή να σχολιάσετε κάποιες από τις παρατηρήσεις του κυρίου Σβάπ. Απλώς για να πω ότι όλα αυτά είναι σωστά. Έχουμε μονάχα γενικές ε, προτάσεις αυτή τη στιγμή, επιτάπητος, και θα πρέπει να επανέλθουμε στα πιο συγκεκριμένα στοιχεία μόνο από τη στιγμή που έχουμε τις ε, οριστικές δημοσιονομικές προοπτικές πολιετής και τις προτάσεις της Κομισιόν τότε μπορούμε να τις εξετάσουμε και να δούμε τι πραγματικές αλλαγέ θέλουμε να θεσπίσουμε. Εγώ προσβλέπω λοιπόν σε μια πολύ καλή συνεργασία με τα μέλη της Επιτροπής μας. Ναι. Θα μπορούσαμε για την άλλη εβδομάδα να έχουμε και ένα προϋπολογισμό πολιετή. Θα δούμε τώρα ποια είναι η θέση των άλλων πολιτικών ομάδων. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε να μας παρουσιάσετε το θέμα αυτό, γιατί ξέρω ότι είσαστε περιζήτη και σε άλλες επιτροπές και εμείς σίγουρα είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί σας και να σας υποστηρίξουμε. Δεν ξέρω τώρα ο κύριο Φαπ θα δώσει τη σκητάλη σε κάποιον άλλο, αλλά ευχαριστώ Άντερς για την παρουσίαση και την εργασία που έχει φέρει σε πέρας. Πάμε στο επόμενο. Είναι πολύ μορφό το πρόγραμμά μας αυτό το απόγευμα. Έχουμε μια γνωμοδότηση την οποία συντάσσομεν για την Επιτροπή Ενέργειας Έρευνας και Βιομηχανίας για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Έχουμε την ανακοίνωση της Κομισιόν από το Δεκέμβριο, έχουμε καθυστερήσει να επιληφθούμε, αλλά ήταν μια σημαντική ανακοίνωση για να λειτουργεί καλύτερα η εσωτερική αγορά ενέργειας. Και όσοι έχετε παρακολουθήσει το έργο της Επιτροπής μας, ξέρετε ότι εδώ και πολλά χρόνια εμείς έχουμε εστιάσει ιδιαίτερα στα δικαιώματα των καταναλωτών στην αγορά ενέργειας. Έχουμε εργαστεί για μια χάρτα καταναλωτή στα θέματα αυτά της ε, ενέργειας και πιστεύω ότι και ο κύριος Κουρέι Αντεκάμπους θα το αντιμετωπίσει αυτό το θέμα, όπως και τη λειτουργία των αγορών σε ό,τι αφορά τα θέματα ενέργειας. Είναι θετικό λοιπόν που θα γίνει αυτή η έκθεση για αυτό το θέμα καθηγητά Κορέη Αντικάμπους, εσείς είσαστε ο εισηγητής για το θέμα αυτό, σας δίνω το λόγο και στη συνέχεια ο κύριος Σφάπ και ο κύριος Μάντες είναι εισηγητές, ο κύριος Κρόσπεκ θα αντικαταστήσει τον κύριο Μάντες. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιοι άλλοι σκιώδεις εισηγητές, εγώ θα πω κάποια λόγια εξ της ομάδας μου, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα είμαι στην πράξη ως σκιώδης εισηγητής και φαντάζομαι ότι έχουμε και κάποιον από την Κομισιόν ή όχι. Δεν βλέπω. Εάν έρθουν θα τους δώσουμε το λόγο. Ας ακούσουμε λοιπόν την άποψη του κυρίου Κουρέι Ντικάμψ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία αυτού του κειμένου, αυτού του νομοθετήματος. Παραμένουν ακόμα πολλά εμπόδια τα οποία δεν επιτρέπουν την πλήρη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς για την ενέργεια. Καταρχήν έχουμε την καθυστέρηση των, ε, της μεταγραφής των οδηγιών και έχουμε φυσικά και φυσικά εμπόδια σε ό,τι αφορά την ε, ε, διασύνδεση των ενεργειακών πόρων μέσα στην Ευρώπη και πολλές φορές η ευθύνη γι' αυτό αφήνεται από τα εθνικά κράτη στους εθνικούς φορείς ενέργειας οι οποίοι έχουν σαν κύριο συμφέρον και κύριο κίνητρο τη διατήρηση του μεριδίου της αγοράς. Υπάρχουν επίσης και εμπόδια που προέρχονται από διαφορετικές ρυθμίσεις ε, για την ενέργεια που εμποδίσουν την είσοδο νέων φορέων στον τομέα αυτό. Παρά τον στόχο λοιπόν για την ενοποίηση της αγοράς εξακολουθεί να ισχύει ο εθνικός κατακαιρματισμός για τις αγορές ενέργειας. Υπάρχουν διάφορε γραμμέ δράση που μπορούμε να ακολουθήσουμε για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά. Πρώτα απ' όλα η επιτάχυνση τη εφαρμογή και υλοποίηση του τρίτου ενεργειακού πακέτου, <clears throat> που σημαίνει και την αποδεσμοποίηση τη παραγωγή διανομή και διανομή ενέργεια. Επίση, την εξασφάλιση μεγαλύτερη διαφάνεια που πρέπει να περιλαμβάνει και το τομέα τη παραγωγή και το τομέα τη διανομή. Υπάρχουν επίση και άλλοι τομεί οι οποίοι προ καλούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό όπως οι ρυθμιζόμενες τιμές, οι επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα και την πυρηνική ενέργεια και οι διαφορές που υπάρχουν για την υποστήριξη της εφαρμογής ανανεώσιμων ενεργειών. Επίσης υπάρχει και ένα ιστορικό πλεονέκτημα των φορέων που είναι ήδη μέσα στην αγορά που εμποδίζει την πραγματική εφαρμογή ε, του ελεύθερου ανταγωνισμού στον τομέα ενέργειας. Επίσης χρειάζεται να υπάρξουν και ρυθμίσεις που θα εξασφαλίσουν την καλύτερη ολοκλήρωση, την συγχώνευση επιχειρήσεων, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη απόδοση σε σχέση με το κόστος σε ευρύτερο επίπεδο από το εθνικό. Αυτό αφορά και τις υποδομές Μεταφορά ενέργεια μεταξύ κρατών μελών και ελπίζουμε ότι εδώ θα υπάρξει το ταχύτερο δυνατό η έγκριση του κανονισμού για τι ενεργειακέ υποδομέ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη συνέχεια θα υπάρξει η ταχεία εφαρμογή του για να μπορέσουν να αρθούν τα φυσικά εμπόδια τα οποία υπάρχουν ακόμα για τη διασύνδεση των κρατών μελών να αντιμετωπιστούν επίση μέσω αυτού και τα θέματα απομόνωση ορισμένων περιοχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική η, η απειλή που προκύπτει από τη μείωση στο μισό περίπου των πόρων που αφορούν την ε, διευκόλυνση Connecting Europe για την ενέργεια, αυτό θα επηρεάσει την εκκίνηση σχεδίων που έχουν να κάνουν με την ε, ενέργεια και την ασφάλεια ενέργειας σε περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν υπάρχει άμεση κερδοφορία σε οικονομικό επίπεδο. Αυξάνονται συνέχεια οι τιμές ενέργειας στην Ευρώπη και αυτό θα συνεχίσει ως τάση για πολύ καιρό. Είναι απαραίτητο λοιπόν να εξασφαλίσουμε προ το συμφέρον του καταναλωτή ότι θα λειτουργήσει η ενεργειακή ε, ενιαία αγορά και για τι επιχειρήσει και για τον καταναλωτή. Είναι απαραίτητο ο καταναλωτή να μπορεί να επιλέγει τον πάροχο ενέργεια με έναν τρόπο ελεύθερο, καλά πληροφορημένο, πληροφορημένο και διάφανο. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει και πλήρη δυνατότητα επιλογής από πολλούς παρόχους. Η τιμή του ηλεκτρισμού ε, σε επίπεδο χονδρικής στα κράτη-μέλη έχει αυξηθεί πιο αργά από ότι η τιμή του ηλεκτρισμού για τον ε, τελικό καταναλωτή, τον ε, ιδιώτη. Πρέπει λοιπόν να αντανακλάτε καλύτερα αυτό στο τελικό λογαριασμό που πληρώνει ο καταναλωτής. Εμείς διατηρούμε αυτή τη στιγμή μια κατάσταση πλασματική η οποία δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάντα. Πρέπει να βοηθήσουμε τους μικρούς καταναλωτές και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να υποφελθούν από τις νέες δυνατότητες που τους δίνει η αγορά. Πρέπει να υπάρξει και μια πιο προορατική αντιμετώπιση για τη διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας με τα λεγόμενα ευφύη δίκτυα και επίσης να υπάρξει και δυνατότητα των καταναλωτών να παίζουν το ρόλο μικροπαραγωγών ενέργειας. Είναι επίση απαραίτητο να υπάρξει μεταλαμβάνευση βελτίστων πρακτικών σε ό,τι αφορά τι καινοτόμε ιδέε και μεθόδου που θα εξασφαλίσουν και καλύτερη προστασία του καταναλωτή από τι εταιρείε παροχή ενέργεια. Μια η ενδιαφέρουσα ιδέα είναι το λεγόμενο collective switching, όπου ένας μεγάλος αριθμός καταναλωτών, μεμονωμένων καταναλωτών, μπορούν να συναθριστούν για να αποτελέσουν ε, να διαπραγματευτεί για παροχή ενέργειας σε συλλογικό επίπεδο στη χώρα μου στις τελευταίες δύο εβδομάδες και μόνο. Υπήρξε μια πρωτοβουλία η οποία κατάφερε να συνενώσει 250.000 καταναλωτές ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν σε, μια, σε ένα πληστηριασμό ενέργειας μαζί με άλλε ενέργειε για να πάρουν πιο ανταγωνιστικέ τιμέ. Αυτό λοιπόν είναι μια δυνατότητα και όλα αυτά τα στοιχεία ελπίζω θα μα βοηθήσουν να διατυπώσουμε μια καλή γνωμοδότηση τη Επιτροπή ΙΜΚΟ ενώπιον τη Επιτροπή ενέργεια. Ευχαριστώ πολύ. σα ευχαριστώ. Δείξατε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία και με βέβαια ότι οι συνάδελφοι θα θέλησουν να απαντήσουν. Ο κύριο Σφάπ. Νομίζω είναι επόμενο ομιλητή, και μετά ο κύριο Κρόιτσμαν. Η κυρία Ρούντερ είναι επίση εδώ. Ο κύριο Φάπ, ευχαριστώ. Ναι, αυτή τη φορά όμως όντως ε, είμαι σκιώτης εισηγητής της ομάδας μου και γι' αυτό λοιπόν καλωσορίζω αυτά που μας είπε ο συνάδελφος Κορέρα Κάμπος. Γνωρίζουμε τον ε, καθηγητή Κορέρα Κάμπος και από άλλους τομείς και γι' αυτό είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία θα είναι άριστη. οι ανακοινώσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα της εύρυθμης λειτουργίας της ιστορικής αγοράς ενέργειας ε, καταδεικνύει ποια είναι τα μέτρα αυτά. Είναι λοιπόν σημαντικό να ασχοληθεί η Επιτροπή μας με τα θέματα αυτά, γιατί η ιστορική αγορά της ενέργειας καταδεικνύει με τρόπο υποδειγματικό ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ακόμα οι αγορές ε, μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των πρώην συνόρων, αν θέλετε, μεταξύ των κρατών μελών. Άρα, καλωσορίζω το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει διαδικασίε επί παραβάση κατά των κρατών μελών που δεν έχουν κάνει σωστή εφαρμογή των σχετικών νομοθεσιών, γιατί παρεμποδίζεται η σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η κυρία Ρέντινγκ υπολόγισε ότι χάνουμε 2,3 δισεκατομμύρια κάθε έτος σε ό,τι αφορά θέματα ψηφιακής ε, τεχνολογίας. Νομίζω ότι παρόμοια είναι τα ποσά και στον τομέα της ενέργειας. Καλώς ορίζω κατά δεύτερον την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ότι σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό τομέα θέλει να εφαρμόσει ιδιαίτερο στα θέματα ανταγωνισμού και βλέπουμε στην Ευρώπη ότι δεν είναι υπερβολικό το μερίδιο της αγοράς αυτής, αλλά είναι ότι είναι πολύ μικρή, πολύ μικρό το μερίδιο του ανταγωνισμού μεταξύ ε, των κρατών μελών και αυτό συνεπάγεται κόστος για τους πολίτες, τους καταναλωτές και δεν ε, συνεπάγεται και την ασφάλεια που θα θέλαμε σε ό,τι αφορά την ανάθεση συμβάσεων, σε ό,τι αφορά και το δευτερογενές ε, δίκαιο. Τα θέματα είναι λιγότερα δύσκολα σε ό,τι αφορά θέματα ενέργειας από τις άλλους τομείς στην Ένωση. Ανακύπτει και το ερώτημα των ρυθμισμένων τιμών. Λίγα είναι τα κράτη-μέλη αυτά, αλλά υπάρχουν κράτη-μέλη στην Ευρώπη που έχουν ορισμένες τιμές και σε ό,τι αφορά το αποκλειστικό δικαίωμα του άρθρου 106 είναι συμβατό προς τη συνθήκη, αλλά σε μια ενιαία αγορά ανακύπτει το ερώτημα κατά πόσον μπορούν να υπάρχουν τέτοιε ρυθμίσει, σε ό,τι αφορά την προστασία του καταναλωτή πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Καλώς ορίζω τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να γίνει ανταλλαγή απόψεων για σημαντικά θέματα σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των τιμών, τη διαφάνεια στις τιμές. Πρόκειται για θέματα τα οποία πλήττουν τους καταναλωτές στις διασυνοριακές περιοχές, επειδή δεν υπάρχει διασυνοριακή διαμόρφωση της αγοράς. Αλλά θεωρώ ότι αυτά δεν αρκούν από μόνα τους και θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα το σημείο αυτό, γι' αυτό λοιπόν θα κλείσω στο σημείο αυτό. Okay. Uh, thank you. Ευχαριστώ πολύ. Όλα αυτά ήταν πολύ σημαντικά. Νομίζω ότι και οι άλλοι συνάδελφοι θα ενημερωθούν. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Κρόιτσμαν, να καλωσορίσω τον κύριο τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εσωτερική αγορά. Θα του δώσω το λόγο σε λίγο, αφού ακούσουμε το σύνολο των σκιωδών εισηγητών. Ο κ. Κρότσμαν έχει στήσει το λόγο. Χωρίς μικρόφωνο, κ. Κρότσμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς έχει ένα σημαντικό καθήκον σε σχέση με την επίτευξη της ε, ευρωπαϊκής ε, αγοράς ενέργειας. Η επίτευξη αυτής της ενοποίησης θα οδηγήσει σε σημαντικά πλεονεκτήματα και για τους καταναλωτές και για τις εταιρείες. Ο καθηγητής ε, ε, Κορέα Κάμπους, τόνισε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές οι οποίοι μπορούν να εξασφαλίσουν και τη δική τους παραγωγή ενέργειας εν μέρη και έτσι να εξαρτώνται λιγότερα από τους παρόχους. Αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε αλλά βλέπουμε ότι στα κράτη-μέλη υπάρχουν διαφορετικές αντιμετωπίσεις για την ιδιωτική παραγωγή ενέργειας. Η Γερμανία από την, ε, με βασίζεται στις ανανεώσιμες ενέργειες, όταν η Γαλλία βασίζεται περισσότερο στην πυρηνική ενέργεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρει ότι μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικέ εξοικονομήσει με μια κοινή προσέγγιση και γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να δώσουμε τη δυνατότητα η ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργεια να γίνει πραγματικότητα. Θα μιλήσω τώρα στα αγγλικά. Γιατί ο αρμόδιο συνάδελφο, ο κύριο Μάντερ, μου τα έγραψε στα αγγλικά. Ευχαριστεί την Κομισιόν για την ανακοίνωση αυτή και τονίζει ότι είναι πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν. Υποστηρίζει ένα κλίμα το οποίο είναι ασφαλές και ανταγωνιστικό για τα ενεργειακά συστήματα. Επίσης, στον τομέα της εφαρμογής θέλει να τονίσει τα θέματα της διασύνδεσης για την εσωτερική αγορά. Μόνο με σωστέ ενεργειακέ διασυνδέσεις μπορούμε να έχουμε ένα υγιή ανταγωνισμό. Ο κ. λοιπόν υποστηρίζει μια ε, επέκταση της χρήσης των υποδομών χωρίς διακρίσεις και επίσης την ενθάρρυνση της καλύτερης χρήσης των δικτύων και τον εξυγχρονισμό τους. Γι' αυτό θα πρέπει να διαρευνήσουμε πιο ε, καινοτόμες ε, προσεγγίσεις και επίσης θα πρέπει να περατωθεί η ενεργειακή από, ε, σε ορισμένων κρατών από το ευρωπαϊκό δίκτυο. Και επίσης πρέπει να εξασφαλιστεί η ολοκλήρωση του συστήματος ενέργειας μέχρι το 2014. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κρόσου. Και τον κύριο Βάντες. Η κυρία Ρούλα έχει το λόγο τώρα. Και εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Νομίζω ότι ο κύριο Κούρια Ελεκάμπους έστειλε τα σωστά μηνύματα. Εγώ υπογραμμίζω ιδιαίτερα και χαιρετίζω το γεγονός ότι η ιδιοπαραγωγή ενέργειας και η αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από όλα τα κράτη και να καταρτιστούν οι κατάλληλες στρατηγικές και να μην αφορά μονάχα τις ίδιες επιχειρήσεις αλλά και τον απλό καταναλωτή. Πρέπει φυσικά να εξασφαλίσουμε μέσα στο πλαίσιο αυτό και την ασφάλεια εφοδιασμού τη ενέργεια. Θέλω να ευχαριστήσω επίση και τον ε, Άντε Φαμ. Νομίζω ότι οι κατευθύνσεις που έχει προσφέρει συμπληρώνουν αυτά τα οποία έχει αναφέρει ο κύριος Κουρέα Αντακάμπος και νομίζω ότι αυτό θα μας οδηγήσουν σε μια καλή γνωμοδότηση. Να κάνω και εγώ κάποια σχόλια συμμετείχα σε και, ένα, σε ένα ενδιαφέρον ε, συνέδριο στο Βερολίνο τον προηγούμενο Σαββατοκύριακο και θα ξέρουν οι Γερμανοί συνάδελφοι ότι η γερμανική πολιτική σε ό,τι αφορά την ενέργεια βρίσκεται σε μια πολύ ενδιαφέρουσα μεταβατική φάση. Να πω δύο λόγια όμως και θεωρώ ότι ε, βελτιώνουμε τελικά την κατάσταση για τον καταναλωτή ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην παρούσα φάση και το ανέφερε αυτό και η Επιτροπή στο σχετικό έγγραφο είναι η έλλειψη ρευστότητας στην ενεργειακή αγορά επειδή δεν είναι ανοιχτές οι αγορές και επειδή υπάρχει μεγάλος έλεγχος από πλευράς των παρόχων όσοι ανταγωνιστές θέλουν να επισέλθουν στην αγορά και να κάνουν προσφορά σε ό,τι αφορά την παροχή ενέργειας δεν έχουν πρόσβαση στις αγορές και γι' αυτό οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν κατά πόσον έχουν τέτοια δικαιώματα δεν γνωρίζουν τι ακριβώς είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πώς μπορούν να τις χρησιμοποιούν. Και το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, αναφέρει ότι θα αναλυφθούν διαδικασίε επί παραβάση κατά των κρατών μελών που δεν έχουν εφαρμόσει τη σχετική νομοθεσία. Κάτι άλλο τώρα που ανέφεραν οι συνάδελφοι. Πώς θα δώσουμε τα σωστά κίνητρα για την ανανέωση των συστημάτων παροχής και για την αποθήκευση της ενέργειας. Αυτό είναι πραγματικά εκ των ουκάνευ. Αν θέλουμε να υπάρχει ε, μια μετάβαση προς τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Θα πρέπει να υπάρχει αποθηκευτικό χώρος, γιατί το ένα δεν μπορεί να υπάρξει χωρί το άλλο. Θα πρέπει να βρούμε τρόπου, λοιπόν, για να διασφαλίσουμε την παροχή κινήτρων για σχετικές επενδύσεις. Και επίσης τίθεται το πολύ ενδιαφέρον θέμα τη διασυνδεσιμότητα μεταξύ των αγορών. Ιδιαίτερος ε, επειδή οι μορφέ πηγής ενέργεια ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η αιωλική, η υδροηλεκτρική, δεν βρίσκονται απαραίτητα στα μέρη όπου χρειάζεται η υδροηλεκτρικη δεν βρισκονται αυτή. Όλα αυτά λοιπόν είναι ερωτήματα τα οποία είναι πάρα πολύ βασικά για την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θεωρώ ότι η αγορά δεν λειτουργεί με επιτυχία σε ό,τι αφορά την παροχή σαφών κινήτρων προς τους επενδυτές. Και διάφορα κράτη-μέλη και το δικό μου κράτος μέλος προσπαθούν να εφαρμόσουν τιμές ε, με οροφή σε ό,τι αφορά την παροχή ενέργειας. Και αυτό φυσικά αντιτίθεται στην αρχή της ανοιχτής αγοράς. Και τέλος, να μην ξεχνάμε τα θέματα λειτουργίας του συστήματος ανταλλαγής ε, ρήπων που δεν εφαρμόζονται και υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και πάλι λοιπόν αυτό παρεμποδίζει τις επενδύσεις. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι θα πρέπει να οριστεί, υπάρχει μάλλον η στρατηγική αλλά δεν εφαρμόζεται σωστά και έτσι προκαλείται αβεβαιότητα. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει σημαντικές αποφάσεις για την σωστή λειτουργία της αγοράς. Αυτό συνεπάγεται ότι από πλευρά μας θα πρέπει και ο καταναλωτής να καταστεί δραστήριος στην αγορά. Αλλά προκειμένου να γίνει αυτό, θα πρέπει να γνωρίζει τι δυνατότητες έχει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εστιαστούμε σε θέματα παροχής. Μάλιστα. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ξέρω αν θα θέλετε να μας διαφωτίσετε. για τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας. Ναι, τώρα έχουν έρθει και άλλοι συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον που εκφράσατε και για την ανακοίνωση αυτή, στην οποία, για την οποία θα θέλαμε να συνεργαστούμε μαζί σας. Συμφωνούμε με τον απότερο στόχο της ολοκλήρωσης ε, της ενεργειακής αγοράς. Σας ευχαριστώ πολύ. Right. Καλώς. Θα αναμένουμε τη συνεργασία μας μαζί σας. Κύριε Ντεκάμπος, θέλετε να μας, να μας επιβεβαιώσετε για το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει καμία διαφωνία από αυτά τα, τα οποία άκουσα από τους συναδελφούς Αυτές οι αναταραχές που έχουμε γνωρίσει τον τελευταίο χρόνο μέσα στα πλαίσια των συζητήσεων για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, δίκτυα ήταν θετική όχι μονάχα για το τελικό αποτέλεσμα που ελπίζω θα, θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα ή τουλάχιστον μέσα στο μήνα αυτό, αλλά ήταν πολύ θετικό γιατί συνεισέφερε νέες ιδέες και οδήγησε σε μια επιτάχυνση των διαδικασιών λόγω παράβασης εναντίον των χωρών που δεν είχαν ακόμα το περιεχόμενο της οδηγίας για τα θέματα αυτά. Είναι πολύ θετικό λοιπόν ότι έχει υπάρξει αυτή η προσπάθεια. Η ευθύνη τώρα της δική μας Επιτροπής είναι πολύ σημαντική σχετικά. Είναι μια ευθύνη σαφής γιατί δεν είμαστε βέβαια η επί της αρμόδια επιτροπή αλλά μπορούμε να παίξουμε σημαντικό ρόλο γιατί τα θέματα αυτά περιλαμβάνονται στη δεύτερη πράξη για την ενιαία αγορά και έχουμε μια απόλυτη νομιμοποίηση για να έχουμε μια στεναρή γνωμοδότηση. Όπως είπε ο κύριος Σφαμπ, δεν είναι μια τυχαία αγορά. Οι ταρίφες στις μεθοριακές ζώνες δεν είναι τέτοιες που να βοηθούν τους καταναλωτές που είναι κοντά σε μια χώρα που είναι φτηνότερη εξακολουθούν οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης να λειτουργούν ως νησίδες ελεγχόμενες όχι από τις κυβερνήσεις αλλά απλώς από τις εταιρείες διανομής ενέργειας. Υπάρχουν χώρες που έχουν κάνει μια τυπική διαδικασία αποδεσμοποίησης αλλά όπου οι διανομής ενέργειας είναι ουσιαστικά ε, από τους παραγωγούς ενέργειας και υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες εξακολουθούν να στρεβλώνουν τις ε, τιμές και τα τιμολόγια με επιδοτήσεις και άλλε ενέργειες που είναι εμπόδια για την είσοδο άλλων παροχών. παρόχων. Οι τιμές είναι ψηλέ και ξέρουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσουν να αυξάνουν μέχρι το 2030. Γιατί χρειάζεται μια τεράστια προσπάθεια εξυγχρονισμού στα δίκτυα ενέργειας. Τα δίκτυα είναι πεπαλαιωμένα. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί νέα ισορροπία στα δίκτυα, η αλλαγή της χρήσης ποινική ενέργειας δημιουργεί πολύ νέα, πολλά νέα προβλήματα. Οι ανανεώσιμες ενέργειες έχουν προχωρήσει πολύ περισσότερο τα τελευταία 10 χρόνια από τα προηγούμενα 50 χρόνια, αλλά αυτές οι ανανεώσιμες ενέργειες θα πρέπει να συμβατοποιηθούν με τα δίκτυα διανομής γιατί οι ανανεώσιμες ενέργειες δεν έχουν σταθερή παροχή ενέργειας αλλά διακειμενόμενη. Όσο μπορέσουμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ρευστότητα σε αυτή την αγορά, τόσο μικρότερη αύξηση τιμών θα έχουμε και καλύτερα έλεγχο θα έχουμε και τελικά τόσο το περισσότερο θα επωφεληθούν οι καταναλωτές. Είναι μια μεγάλη πρόκληση τα smart grids, grids τα εφηδίκτια. Το να περιμένουμε θα το λύσουμε το πρόβλημα αυτό μέχρι το 2014 είναι μια εκδήλωση αισιοδοξία που τη χαιρετίζω, αλλά δεν ξέρω αν είναι ρεαλιστική ο κανονισμός μας για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας ενεκρίθη τον, έπρεπε να εκριθεί τον Ιανουάριο, τώρα είναι Μάρτιος και δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό και τον επόμενο μήνα. Υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά τα εμπόδια τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και τέλος, σε σχέση με αυτά τα οποία είπε ο πρόεδρος Χάρμπορ για τη συνδιάσκεψη στο Βερολίνο, νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο γνωρίζω πολύ καλά. Τα κίνητρα για την ανακαίνιση του δικτύου διανομής και ε, αποθήκευσης ενέργειας του προγράμματος Connecting Europe είναι τώρα 5 δισεκατομμύρια ενώ ήταν 9,9 στο αρχικό πρόγραμμα της Κομισιόν. 5 δισεκατομμύρια είναι πολύ λίγα πρέπει να χρησιμοποιηθούν βέβαια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ακόμα πιο σημαντικό όμως είναι να υπάρξει μια σωστή προσέγγιση για την μεταρρύθμιση της αγοράς. Η μεταρρύθμιση της αγοράς μπορεί να γίνει με την ε, προτυποποίηση, με τους μηχανισμούς που θα εξασφαλίσουν το συντονισμό και τη συμβατότητα των δικτύων των εθνικών στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και εν κατακλείδη ήθελα να σας πω ότι το θέμα αυτό της ενέργειας στην εσωτερική αγορά θα είναι μια καταπληκτική περίπτωση που θα μελετούν οι επιστήμονες και οι ακαδημαϊκοί στο μέλλον. Είναι μια <clears throat> μεγάλη πρόκληση. Αν δεν πάει καλά θα υπάρξει μεγαλύτερη δυσπιστία για την αξία της ε, ενιαίας αγοράς. Αν καταφέρουμε όμως να λειτουργήσει σωστά η ενιαία αγορά της ενέργειας, θα υπάρξει μεγαλύτερος ενθουσιασμός <clears throat> και αισιοδοξία για όλη την Ευρώπη. Υπάρχει λοιπόν και ο συμβολικός χαρακτήρας για τα ενεργειακά θέματα, γιατί είμαστε ενώπιον ενός θέματος που είναι πολύ νευραλγικό και όπου μπορούμε να εξασφαλίσουμε πολλά πλεονεκτήματα. Για το χρονοδιάγραμμα. Το χρονοδιάγραμμα, όπως το έχω προτείνει, είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. Μάλλον, συγγνώμη. Πρέπει 19 Μαρτίου να αποσταλεί το σχέδιο γνωμοδότησης το σχέδιο 12 ε, ναι, Απριλίου θα γίνει η συζήτηση και 25 Απριλίου η προθεσμία <clears throat> για τις τροπολογίες. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε λοιπόν να καλύψουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ. No, I'm sure you're right. Σίγουρα θα το πετύχουμε. Μέχρι τις 29 Μαΐου θα πρέπει να υιοθετήσουμε την πρότασή μας. 30 Μαΐου είναι η τελική προθεσμία. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια προσπάθεια και στην Επιτροπή Βιομηχανίας εκ των προτέρων. Ε, καλά κάνετε και μας υπενθυμίζετε τη σημασία που έχει για την εσωτερική αγορά του συγκεκριμένο θέμα, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει σχέση με τους καταναλωτές. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλα θέματα επίσημα για την Επιτροπή. Έχουμε ένα τελικό θέμα το οποίο θα το έχουμε συνεχώς από εδώ και πέρα μέχρι τη στιγμή που θα κλείσουμε όλες τις συζητήσεις ε, νομοθετικού τριμερούς διαλόγου. Όσοι παρακολουθούν τις εργασίες μας γνωρίζουν ότι στην τελευταία συνάντηση οι εισηγητές ανέλαβαν την εντολή να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για κάποια θέματα. Έχουμε και άλλα δύο θέματα τα οποία είναι σε εκκρεμότητα. Θα τα συνδυάσουμε και θα παρουσιάζουμε τα λεγόμενα progress report. Εγώ είμαι ο μόνος εισηγητής για να θέσετε τις ερωτήσεις σας, αλλά θα παρουσιάσω τις εκθέσεις και εκ μέρους της κυρίας ε, Ρόιτεβα και εκ μέρους της κυρίας Λεγκρίπ για διαφορετικά θέματα. Και αν θέλετε να θέσετε ερωτήσεις μπορείτε να το κάνετε μεν. Αλλά αυτά τα οποία θα πω ελπίζω να βοηθήσουν έτσι ώστε όλοι να είναι ενήμεροι για την πρόοδο του διαλόγου αυτού του τριμερούς και να διασφαλίσουμε τις διαπραγματεύσεις, την διαφάνεια των διαπραγματεύσεων. Βέβαια ξέρετε ότι ό,τι συζητιέται στην ε, συνάντηση αυτή ε, δεν δημοσιεύεται, αλλά μπορούμε παρόλα αυτά να σας ενημερώνουμε. Καταρχάς, το πακέτο ευθυγράμμισης της νέας νομοθετικής πρωτοβουλία. Όσοι είστε ενθουσιασμένοι με τις προσπάθειες γυρνίασης της εσωτερικής νομοθεσίας, ξέρετε ότι είναι κάποια μέτρα τα οποία έχουν σαν στόχο ε, κάποιες ρυθμίσεις τεχνικής φύσεως για την εποπτεία της αγοράς και κάποια άλλα θέματα που αφορούν την εφαρμογή των μέτρων αυτών και την αποτελεσματικότητα των προτάσεων αυτών. Η κυρία Ρόιτεβα είναι η συγγήτρια, η οποία ασχολείται με εννέα διαφορετικές οδηγίες με εντελώς διαφορετικά θέματα. Υπάρχουν ένα-δύο επιπλέον στοιχεία, ιδιαίτερα τεχνικά, τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Είχαμε λοιπόν ένα τριμερή διάλογο στις 5 Δεκεμβρίου. Υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες σε όλα αυτά τα θέματα και άλλωστε και στόχος ακριβώς αυτών των ρυθμίσεων μέσα από τις οποίες λειτουργούν οι ομάδες εργασίας του Συμβουλίου είναι οι λεπτομέρειες οι οποίες επηρεάζουν ε, την εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων. Υπάρχουν ε, λοιπόν πάρα πολλές τεχνικές προσπάθειες που γίνονται σε επίπεδο διαδρόμων θα έλεγα σε αυτή τη φάση έτσι ώστε να καταλήξουμε επίσημα στις τελικές ρυθμίσεις. Από τότε που ξεκίνησε ο διάλογος έχουν υπάρξει πολλές συναντήσεις ανάμεσά μας και τους εκπροσώπους των κρατών μελών στο Συμβούλιο. Έχει υπάρξει κάποια πρόεδρος και κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας και τώρα κατά τη διάρκεια της Ιρλανδικής Προεδρίας να υπενθυμίσουν συναδέλφους ότι κάθε έξι μήνες αλλάζει η Προεδρία των Ομάδων Εργασίας του Συμβουλίου. Υπάρχουν τεχνικές ρυθμίσεις για την ένταση τους λεγόμενους εντατήρες ή προεντατήρες των ζωνών ασφαλείας των αυτοκινήτων και τους μηχανισμούς ε, ε, θέσης σε λειτουργίας των ε, αερόσακων των αυτοκινήτων. Να μην ξεχνάμε επίσης και το θέμα του χρονοδιαγράμματος. Η συγκήτρια συνεργάζεται με την Επιτροπή και το Συμβούλιο για να γίνουν σεβαστά τα χρονοδιαγράμματα Έχουμε μία επιπλέον συνάντηση αυτή τη βδομάδα σε δύο μέρες στις 6 του μηνός. Θα έχουμε επίσης και στις 19 Μαρτίου μία συνάντηση σχετικά με ε, τις αντίστοιχες οδηγίες και η τελική θέση ε, θα τεθεί ε, προς έγκριση από πλευρά σας στις 11 Απριλίου. Και μετά θα πάμε στην Ολομέλεια. Λοιπόν, εκεί βρισκόμαστε για τα θέματα της κυρίας Ρόιτεβα. Δεν ξέρω αν έχετε ερωτήσει. Όχι. Το επόμενο θέμα είναι η δική μου έκθεση, η δική μου οδηγία μάλλον με την οποία ασχολούμαι. Now those of you who were enthusiasts for this will know that it was actually voted in this committee last summer, uh, but we decided not to. Για τις βιοτεχνίες ε, και τέτοιου είδους ενασχολήσεις έχουν προτείνει κάποια επιμέρους επαγγέλματα όπως τους ε, ναυπηγούς οι οποίοι ε, μερικές φορές δεν καλύπτονται από τις υπάρχουσες ρυθμίσεις και έχει υπάρξει πρόοδο στα κενά τα οποία έχουν σημειωθεί. Έχουμε προκαλέσει μια αρκετά χρήσιμη συζήτηση με τους ναυπηγούς έτσι ώστε να αλλάξουν οι κατηγορίες των σχεδίων πλοίων και τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται για, την, για τον χαρακτηρισμό της, κατα, των, της καταστάσεως στην οποία βρίσκεται ε, η θάλασσα κάθε φορά. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες χρήσιμες προτάσεις που έχουν ακουστεί. Έχουμε προκαλέσει αρκετές συζητήσεις γύρω από τα θέματα αυτά στο Συμβούλιο. Θα περιμένουμε τώρα τις τελικές ε, προτάσεις Έχουμε παρόλα αυτά κάποιες βασικές συμφωνίες για όλες τις αλλαγές που θέλουμε να γίνουν σχετικά με τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Θα υπάρξουν δύο τεχνικές συναντήσεις, στις 6 και στις 25 Μαρτίου και ελπίζουμε να υπάρξει ένας τριμερής διάλογος για τις αρχές Μαΐου. Μέχρι τότε ελπίζω να είμαστε σε θέση να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες συμφωνίες. Δεν ξέρω αν έχετε περισσότερες ερωτήσεις για τα θέματα αυτά. Όχι. Και τώρα έχω και την έκθεση της κυρίας Λεγκρίπ. Θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Σβάμπ. Ξέρω ότι σας έχει ενημερώσει η κυρία Λεγκρίπ, οπότε μπορείτε να ενημερώσετε εσείς αν θέλετε. Όχι εσείς λέει ο κύριος Σβάμπ. Ναι, κοιτάξτε, εγώ έτσι κι αλλιώς προεδρεύω σε όλες αυτές τις συναντήσεις, λέει ο πρόεδρος και συνεχίζει. Η πρώτη τριμερή συνάντηση για τον ενιοποιημένο τελωνιακό κώδικα και το πακέτο ε, κατάθεσης εκ νέου του κώδικα αυτού. Είναι κάτι με το οποίο ασχολείται η κυρία Λεγκρίπ και έχει πάρει συγκεκριμένη εντολή γι' αυτό πριν ένα μήνα. Υπάρχουν κάποια περίπλοκα θέματα γύρω από το συγκεκριμένο θέμα γιατί ε, δεν υπάρχει μεγάλη άνεση χρονική Η προθεσμία για τις προτάσεις αλλαγών είναι ο μήνας Ιούνιος, οπότε πρέπει να βιαστούμε να περάσουμε από την Ολομέλεια γύρω από τον νέο τελωνιακό κώδικα. Πάντως είναι περίπλοκο τεχνικά το θέμα. Υπήρξαν ε, λοιπόν συναντήσεις, η τελευταία ήταν μια τρίωρη χρήσιμη συνάντηση, κάθε θεσμικό όργανο παρουσίασε τις απόψεις του για πρώτη φορά συνολικά και ορίσαμε τα θέματα πάνω στα οποία θα πρέπει να υπάρξει μια κάποια συμφωνία. Το πιο περίπλοκο από τα θέματα που αφορούν τον τελωνιακό κώδικα είναι ότι το βασικό στοιχείο μεταρρύθμισης της πρότασης αυτής είναι η ευθυγράμμιση με τη συνθήκη της Λισαβόνας σχετικά με την εκχώρηση εφαρμοστικών πράξεων και ε, πράξεων ε, εκτελεστικής παραχώρησης που δεν καλύπτονται από τις ρυθμίσεις που ισχύουν σήμερα. Έχει υπάρξει προσπάθεια ως προς αυτό από το Συμβούλιο, αλλά πολλά μένει να γίνουν και θα πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρειες. Ένα από τα θέματα λοιπόν ήταν ε, το να υπάρξει ένα βασικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τις εκτελεστικές πράξεις και τις πράξεις εξουσιοδότησης έτσι ώστε οι πολιτικές μας προτεραιότητες να εκπροσωπούνται και αυτές στα πλαίσια της συγκεκριμένης διαδικασίας. Απαιτείται να υπάρξει μια συγκεκριμένη πρόταση του Κοινοβουλίου για την μεταρρύθμιση του τελωνιακού κώδικα, έτσι ώστε οι προτεραιότητές μας, όπως και οι προτεραιότητες και των άλλων οργάνων, να ισορροπηθούν και να εκπροσωπηθούν σωστά. Υπάρχουν και άλλα θέματα σχετικά ε, με τα θέματα προσωρινής φύλαξης ε, από πλευράς των τελωνιακών αρχών, θέματα πληροφορικής τεχνολογίας, θέματα ελέγχου, θέματα χορήγησης προσωρινών εξαιρέσεων, θέματα προσωρινών ρυθμίσεων, μεταβατικών ρυθμίσεων. Υπάρχουν επίσης και το θέματα τα σχετικά με με την μεταχείριση των επιχειρήσεων στα πλαίσια των τελωνιακών διαδικασιών και επίσης θέματα σχετικά με την δημιουργία συνθήκων για την αμοιβαία αναγνώριση των διαδικασιών. Επίσης για την προέλευση των αγαθών στις τελωνιακές διαδικασίες, θέματα τα οποία είναι κρεμή ακόμα, δεν έχουμε συμφωνήσει με το Συμβούλιο και αυτή είναι μια από τις κύριες δυσκολίες. Χρονικές, ε, ε, χρονικά όρια στα χρέη, και τις οφειλές, ε, αξιολόγηση, εκτίμηση. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα δούμε λεπτομεριακά και ελπίζουμε να προχωρήσουμε σε όλα αυτά τα θέματα. Η κυρία Λεγκρή στην, ε, σύνοψή της καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν, έχουν τους ίδιους στόχους αλλά έχουμε διαφορετικές διατυπώσεις για τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Χρειαζόμαστε τεχνικό έργο για ευθυγραμμίσουμε την ε, προσέγγισή μας. Πιστεύω όμως παρόλα αυτά με τη βοήθεια του Θεού μπορούμε να φτάσουμε την κατάλληλη ποιότητα στην ε, σύνταξη των νομοθετημάτων αυτών ώστε να πετύχουμε τους πολιτικούς μας στόχους. Κάποια από αυτά τα θέματα λοιπόν γίνεται σε τεχνικό επίπεδο, είναι με εξουσιοδότηση χωρίς να αλλάξουμε το πολιτικό πλαίσιο και υπάρχουν και κάποιες σημαντικές διαφωνίες και αποκλήσεις σε κάποια θέματα. Θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε στον κύριο τριγωνικό διάλογο. Προσπαθούμε προς το παρόν να καλύψουμε τα θέματα αυτά τα δύο για να καλύψουμε και το χρονοδιάγραμμα. Κάναμε όμως σαφές προς την Ελλανδική Προεδρία ότι είναι περιορισμένοι οι πόροι μας και σε ό,τι αφορά τη χρονική αλληλουχία αυτών των θεμάτων θα πρέπει να δώσουμε την σωστή χρήση των πόρων μας και με τον τρόπο αυτό άλλα θέματα όπως οι δημόσιες προμήθειες μπορεί να καθυστερήσουν αδειρήτως. Αλλά θα πρέπει τελικά όλα αυτά τα προβλήματα να επιληθούν. Αλλά έτσι είσαστε και πλήρω ενημερωμένοι. Ερωτήματα? Κύριε Σουάπ, όχι, ου. Κυρία Ρούλα, κυρία και σας τα παρούσα. Να σας υποστηρίξω. Θέλω να υποστηρίξω λοιπόν αυτό το οποίο είπατε, ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε σωστά και τη χρονική αλληλουχία αυτών των θεμάτων. Οι μικρές ομάδες βέβαια έχουν ε, δυσκολίες για να μπορούν να συμμετάσχουν σε πάρα πολλές τεχνικές συναντήσεις και δεν μπορούμε σε όλα τα θέματα να παρακολουθήσουμε την κατάσταση, αλλά ε, αυτό που μας ενδιαφέρει πρωτίστως είναι να προχωρήσει σωστά διαδικασία. Εντάξει, δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει να πει κάτι. Good. Well, thank you very much. Εντάξει, σας ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία σας στη σημερινή συνεδρίαση. Η επόμενη συνεδρίασή μας, αν θέλει ο Θεός, θα είναι 20 Μαρτίου Τετάρτη έχουμε συνεδρίαση πρωί και απόγευμα από τις 9 στο 10.30 και από τις 3 ως τις 6.30 και 21 Μαρτίου από τις 9 ως τι 12.30 και από τις 3 ως τις 6.30. Θα ήθελα να ζητήσω από όλα τα πολυπληθή μέλη που είναι εδώ πέρα, αλλά κυρίως να αναφερθώ στους συντονιστές των πολιτικών ομάδων, να εξασφαλίσετε παρακαλώ ότι έχουμε πλήρη παρουσία την Πέμπτη το απόγευμα, γιατί πολλοί κόσμος έχει την τάση να την κάνει την Πέμπτη το απόγευμα. Και όλες αυτές οι ημερομηνίε βρίσκονται στο χρονοδιάγραμμα. Ξέρω ότι όλοι θέλουν να πάρουν σπίτι τους νωρίς το, το Σαββατοκύριακο, αλλά επειδή ξεκινάμε μονάχα την Τετάρτη στις 9 η ώρα, θα έχουμε Δευτέρα και Τρίτη ελεύθερη. Πρέπει να αρχίσουμε να επιταχύνουμε τους ρυθμούς εργασίας μας τώρα που έχουμε αυτές τις ε, συνεδριάσεις που δεν είναι από τρίτη μεσημέρι ω πέμπτη μεσημέρι λόγω περιορισμού ερμηνείας και διερμηνείας, αλλά είναι Τετάρτη και Πέμπτη. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλοι είναι εδώ πέρα παρόντες την Πέμπτη το απόγευμα και κυρίως οι συγητές. Εξασφαλίστε παρακαλώ για τα μέλη της πολιτικής σας ομάδος ότι θα υπάρχει πλήρης προσέλευση και παρουσία και αύριο συνεδριάζουν οι συντονιστές το απόγευμα για να υπάρξει και σχεδιασμός της στρατηγικής μας για το υπόλοιπο τμήμα της θητείας μας, ιδίως σε σχέση με τις πολιτικές πρωτοβουλίες που θέλουμε να αναλάβουμε. Απλώς σας το υπενθυμίζω αυτό λοιπόν στη δημόσια συνεδρίαση. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας, ευχαριστώ και το προσωπικό μας και τους διερμηνείς και θα τα πούμε στις 20 Μαρτίου.